if you don't mind, Paul. Yeah, I'm here. I, but I'm so shy. I, I, <laughs> so hello everybody for our... Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην απόψηνή μας συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω όλους θερμά στην νυχτή συνεδρίαση σε μια ενοποιημένη φορολογική βάση. ορίζω και τους προσκεκλημένους μας. Δύο. Σε λίγο όμως θα τους παρουσιάσουμε. Δύο είναι οι ομάδες συζήτησης, υπάρχει και αίθουσα ακρόασης. Πολλοί μας παρακολουθούν και από το διαδίκτυο. Και καλωσορίζω τον κύριο Βαλιάν Μουταλιέ. από την Τάξουτ που θα λάβει το λόγο πριν από τους τέσσερις κύριους ομιλητές θα μας παρουσιάσει τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε έχει μακρά ιστορία η πρόταση. Είμαι από τους πιο παλιούς εδώ. Πρέπει να είναι η τρίτη μου συζήτηση για εταιρικό φόρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω ορίζω λοιπόν τους δύο συγκεκριτές εδώ. Τάγκ και Λαμασούρ. Θα λάβουν και αυτοί το λόγο ασφαλώ. Δεν κάνω άλλε ανακοινώσει ω πρόεδρο για να δώσω το λόγο στου εισηγητέ και μετά στην Επιτροπή. Το αλλάξαμε πάλι. Ο Δεν είναι εδώ. Α Ας ξεκινήσω ο Άλλα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας που δέχτηκα να γίνει αυτή η δημόσια ανταλλαγή απόψεων. Το είπατε άλλωστε κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, θελήσαμε να ακούσουμε τους ε, εκπροσώπους των βασικών κατηγορίων των stakeholders. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, αλλά επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, τα συνδικάτα και κάποιες μίκιο που ενδιαφέρονται και οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί φορεί σε αυτό το τομέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή, τον κύριο Μουταγή, που τον ευχαριστώ που ήρθε σήμερα. Εντάχει, γνωρίζετε όλοι το θέμα, όλα τα θέματα, ξέρετε τις ανησυχίες μας. Εγώ θα επέμενα επί τριών-τεσσάρων σημείων. Εμπρότης, πρόκειται περί συνεπώς, και η σύνταξη δεν είναι πολύ ακριβή σε κάποια σημεία. Εάν θέλουμε να, έχουμε, να παρουσιάσουμε μια ενότητα παρόλο που έχουμε 27 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, πρέπει να το συζητήσουμε. Από πλευρά επιχειρήσεων ακούμε να λένε ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν έχει ενδιαφέρον παρά μόνο τα δύο κείμενα υιοθετηθούν και κυρίω αν εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Το CCCTB ε, ήμουν εισηγητής, συνεργάζομαι με τον Πολ Τάγκ, που είναι ο εισηγητής του πρώτου κειμένου. Αυτό θεωρούμε εξ αρχής. Θέλω να δούμε τι, θε, θέλουν και τι σκέφτονται οι άλλοι παρεμβαίνονται σήμερα. Θέλουμε το απλούστο δυνατό σύστημα. Αλλά βλέπουμε ότι εφόσον δεν έχουμε εναρμονίσει τα λογιστικά των επιχειρήσεων, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο λογιστικό φορολογικό σύστημα που θα είναι περίπλοκο να εφαρμοστεί. Για το CCCTB ένα βασικό πρόβλημα είναι η κατανομή των φόρων μεταξύ των διαφόρων χωρών, εκεί που ασκούν οι εταιρείε τη δραστηριότητά του. Η προτινόμενη προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εμπνέεται από αυτά που κάνει ο ΣΑ, μήπω αυτή είναι η καλύτερη λύση. Μήπως το να λάβουμε υπόψη τα ώρα, τα, άειλα στοιχεία ενεργητικού ε, δημιουργεί προβλήματα κυρίως για την ψηφιακή οικονομία και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να κάποια από τα βασικά μας ε, ερωτηματικά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πολ Τάγκ είναι άλλος συγγητής. Ε, Πολ, έχεις και εσύ το λόγο. Ευχαριστώ Μάρκους. Μακρά ιστορία. Μας την υπενθυμίσατε. Ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε όμως την ιστορία και θέλουμε αυτή τη φορά να το κάνουμε κάπως διαφορετικά. Το Ευρωκοινοβούλιο σαφέστατα σε έργο της Επιτροπής Τάξη επί την ηγεσία του Αλέων Λαμασούρ στηρίζει την ιδέα υποχρεωτικού του CCCTP. Ε, αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόταση. Η εφαρμογή της προτάσεως ε, μας απασχολεί. Έχουμε και την ενοποίηση που θέλουμε, το τρίτο C του CCCCTB. Θα συνεργαστούμε, Αλένα Μασούρ και εγώ, συνεργαζόμαστε γιατί ανήκουν μαζί όχι μόνο λογικά, τεχνικά, αλλά και πολιτικά. Οπότε θεωρούμε ότι είναι κοινή προσπάθεια και ο λόγος τον οποίο το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την πρόταση εν γέννη σχετίζεται με δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, χρειάζονται ισότιμε συνθήκε για όλου και για τι μεγάλε εταιρείε και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει πληρώνουν ένα τρίτο παραπάνω φόρου από ότι οι μεγάλε εταιρείε. Αυτό γίνεται τώρα. Αλλά δεν θέλουμε μόνο αυτό, τι ισότιμε συνθήκε και έλλειψη στρέβλωση, αλλά θέλουμε να επικρατήσει μια βασική στοιχειώδη δικαιοσύνη. Δύσκολο να καταλάβει κανεί γιατί η μικρότερη εταιρεία θα πληρώνει περισσότερου φόρου από ότι μια μεγάλη. Ταυτόχρονα κάτι δεν άλλαξε, αληθεύει. Έχει και, είναι και βολικό για τις μεγάλες εταιρείες να πληρώνουν σε ένα σημείο επαφής ε, άπαξ τους φόρους που χρωστάνε και όχι σε κάθε κράτος μέρος ξεχωριστά. Αυτές οι προτάσεις ε, έρχονται σε κάποια κρίσιμη περίοδο τι είδαμε, ο Τραμπ πρότεινε να μειώσει το φόρο που επιβάλλει επί των επιχειρήσεων. Σε μία σελίδα το έγραψε αυτό, σε ένα μία σελίδα α4. Αυτό το στυλ χρησιμοποιούν οι λαϊκιστές, βλέπετε. Δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, αυτό που γράφει, αλλά δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες. Αυτή την αλλαγή θα δούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια θα είναι η ευρωπαϊκή απάντηση. Και στη Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit λένε ότι θέλουν να αλλάξουν τους φόρους των επιχειρήσεων. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Θα μπούμε σε αγώνα, κάτωθι, αγώνα, ή θα δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση που στρέφεται κατά αυτού του αγώνα αλλά δημιουργεί ένα παράδειγμα και εντός και εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι ευρύτερο θέμα. Καλό που διεξάγεται αυτή η ακρόαση. Ευχαριστώ και τον προτέρων για τη συνεισφορά των όσων θα μιλήσουν. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα μιας διαδικασίας. Με τα χαράς να ακούσουμε τα όσα έχουν να πούν τα διάφορα μέλη θα μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ, Πολ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομη παρουσίαση της προτάσεως. Βαλέρ Μουταριέ, ο πρώτος, θα μιλήσει. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε συγητέ, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα σχετικά με το ζήτημα της ακράσεως, δηλαδή την κοινή ενωπημένη βάση φορολόγηση των εταιριών. Ο τίτλος αναφερόταν επίσης και στη συνέχεια που δίδεται στις εκθέσεις της ειδική Επιτροπής τάξε 1 και τάξε 2 Θέλω να πω ότι από αυτή την πλευρά δεν έχω πολλά να προσθέσω εν συγκρίση με αυτά που ο Επίτροπος Μοσκοβισή είπε στην Ολομέλεια τον Μάρτιο, εκτός από το εξή ίσως. Η συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στη διαμόρφωση του θεματολογίου για περισσότερη δικαιοσύνη στο ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα και τη μεγαλύτερη ισοτιμία ήταν αποφασιστική σημασίας. Μας επέτρεψε να προχωρήσουμε να προοδεύσουμε ούτω ώστε να μεταμορφώσουμε τις ε, δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε σε διεθνή βήματα και φορείς, να τα μετατρέπουμε σε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το τρόπος αποκτώντας ένα δίκαιο σύστημα, αλλά και μια ασφάλεια δικαίου στον τομέα της φορολόγησης των ε, εμπορευομένων μας διότι αυτά τα δύο στοιχεία θελήσαμε να προωθήσουμε με, το, με τη δέσμη προτάσεων που θέτησε τον Οκτώβριο πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλαμε να έχουμε ένα σύστημα που είναι δικαιότερο, στεναρότερο, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να σταθεροποιήσουν τη φορολογική τους βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και να αποφύγουμε τη διάβρωση της εν λόγω βάσεως, αλλά έχουμε και ένα σύστημα που προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους οικονομικούς φορείς ένα περιβάλλον απλούστερο, φθηνότερο, ανταγωνιστικότερο εντός της ενιαίας αγοράς. Ε, είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση διότι συνεπάγεται τη συνεχή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη συζήτηση και διατηρούμε την όλη ε, ορμή που έχει αποκτήσει το θέμα και θέλουμε μια κοινή υλοποίηση των μέτρων σε αυτό τον τομέα μια στιγμή που ακούγονται εδώ και εκεί διάφορες εκκλήσεις για περισσότερη υποστήριξη της ασφαλείας δικαίου περισσότερο αυτό παρά να έχουμε ένα δίκαιο σύστημα ε, φορολόγησης των επιχειρήσεων. Ε, η πρόταση που έχουμε υποβάλει πέρσι τον Οκτώβριο προσπαθεί να ακολουθήσει τους δύο αυτούς στόχους, να προσπαθήσει να τους πετύχει. Σε σχέση με την αρχική πρόταση του 2011, ενσωματώνει όλο το διατακτικό, επιτρέποντας έτσι την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εντός εσωτερικής αγοράς, διότι νέα αυτή η πρόταση ενισχύθηκε σημαντικά όσον αφορά τις διατάξεις ε, καταπολεμήσεως των καταχρήσεων και προσφέρει όπως και το 2011 το ίδιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις κυρίως όσον αφορά τη μείωση του διοικητικού κόστους και τη δυνατότητα να κινούνται και εκτός των εσωτερικών συνόρων με πιο χαμηλό κόστος και να σέβονται τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φορολογία των επιχειρήσεων. Το νέο σύστημα που προτείναμε θεσπίζει επίσης και διάφορα στοιχεία που επιτρέπουν να προσφέρουμε σε επιχειρήσεις ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό πλαίσιο. Έχουμε τρία καινούργια στοιχεία που έχουμε θεσπίσει αυτό το πλαίσιο, πολύ σημαντικά. Το πρώτο, ένα σύστημα φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό εδράζεται επί αναλύσεως των παρόντων συστημάτων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίζεται επί του συστήματος που θεωρήθηκε το πιο αποδοτικό στο τέλος ανάλυσης, δηλαδή μία μεγάλη μείωση του κόστους έρευνας και ανάπτυξης, δεύτερος μηχανισμός που εντάσσεται ευνοεί τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τα ίδια κεφάλαια και όχι μέσω χρεώσεως αυτών, επιτρέπει ε, μια ουδέτερη φορολογική αντιμετώπιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση και το μέσω δανείων και το κεφαλαίων. Και τρίτον, μετά την ανάλυση που κάναμε, πριν την ενοποίηση των δύο κειμένων, ε, προσφέρουμε ένα μηχανισμό αντιστάθμισης των διασυνοριακών απολειών. Προς και στο δεύτερο στάδιο της προτάσεως θα έχουμε τα πραγματικά ωφέλη και τα κέρδη που επιτρέπει το στάδιο αυτό την ενοποίηση εντός της εσωτερικής αγοράς των μέτρων να επενθυμίσω το πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει, επιθυμεί διακαώς το σχέδιο αυτό που περιέγραψε ο κύριος Λαμασούρ να πετύχει τον απότερο στόχο, το δεύτερο στάδιο με την διότι αυτό το στάδιο δίνει και τα περισσότερα κέρδη. Με τα χαράς να ακούσω τις ε, απόψεις των ε, μελών του πάνελ της απογευματινής ακροάσεως μας και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του που είναι συνεχής όσον αφορά προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη πιο ανταγωνιστικής και δίκαιης φορολόγησης των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή. Και τώρα καλωσορίζουμε το πρώτο πάνελ. James Watson από την Business Europe. Gergat Humer και Olivier Μπουταλιτάφτ από την Accountancy Europe. Αυτή τη σειρά θα ακολουθήσουμε. Ο καθένας έχει πέντε λεπτά. Ο James Watson, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την πρόσκλησή της. Να αρχίσουμε το CCTB, μια που έχουμε ακόμη την ευκαιρία να δούμε τα θέματα της φοροαποφυγής κάπου λίγο πιο αργά πρώτα πρώτα αυτή η έννοια που συζητούμε βελτιώνει η νέα αγορά και βοηθά επενδύσεις και απασχόληση και διασυνοριακά. Η επιχείρηση, Τουρκία ένα μόνο κράτος μέλος, θέλει να επεκταθεί σε μια άλλη αγορά. Ε, φανταστείτε ότι ο κίνδυνος της επέκτασης στην νέα αγορά θα μειωθεί κατά πάρα πολύ. Αν το ξέρει ότι πρόκειται να έχει ζημία εκεί και μπορεί να το αντισταθμίσει με τα κέρδη στην χώρα προέλευσης. Οπότε βλέπουμε ποια είναι τα υπέρ της υπόθεσης βεβαίως και το CCTV πρόκειται να οδηγήσει και σε ανάλογες τιμολογικές πολιτικές σε σχέση με την φορολόγηση. Πέραν αυτών, ο κύριο Λαμασούρ μας είπε όσον αφορά την ενωπημένη βάση φορολογίας ότι θα υπάρχει μία βάση που μπορεί να μην ωφελεί το περιβάλλον το επιχειρησιακό. Ε, αμοιώσει το διοικητικό κόστος. Μπορεί αυτό να βοηθήσει την κοινή βάση και έτσι να υπάρχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε έχουμε τους διάφορους κανόνες εδώ, CFC και κάποιους περιορισμούς όσον αφορά το κατά πόσο μπορούν να εκπέσουν οι απώλειες και άλλα κόστη των επιχειρήσεων. Τώρα, όσον αφορά αυτή την πρόταση για το CCCTV και την ε, ενοποίηση, νομίζω ότι πολλές επιχειρήσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η πρόταση. Ε, νομίζω ότι όλες θεωρούν ότι μπορεί αυτό να προχωρήσει, ούτω ώστε έτσι να υποστηριχθεί περισσότερο η ανταγωνιστικότητα. Τώρα για να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα θέματα. Ε, υπάρχει ο φόβος ότι έτσι δεν θα υπάρχει ευελιξία σε διάφορα κράτη-μέλη από την πρόταση για το CCCTB δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η παγκόσμια οικονομία ή το φορολογικό περιβάλλον. Οπότε αυτό θα δυσκολέψει την ομοφωνία στο Συμβουλίο. Θα είναι δύσκολο να προσαρμοστεί το CCTB σε σχέση με τις προαναφερθήσεις αλλαγές. Επίσης ξέρουμε ότι κάποιοι θα είναι χαμένοι και κάποιοι κερδισμένοι σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης υπάρχει ο φόβος ότι κάποιοι που θα χάσουν σε φορολογικά εταιρικά έσοδα θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν τα απολεσθέντα με την αύξηση συντελεστών. Οπότε θα υπάρξει αύξηση, ιδίως στα κράτη-μέλη, αύξηση των φόρων. Επίσης, άλλο, άλλη μέρη, άλλος φόβος, σε σχέση με τις μεταβλήσεις ότι και έκλειδα κατανομής ε, και τα σχετικά με τις επενδύσεις θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα πρότυπα, τα επιχειρηματικά, όπως το είπε ο κύριος Λαμασούρ. Εάν υπάρχουν κάποιες επενδύσεις χειροπιαστές. Καλά τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα διατυπώνει, αλλά αυτού του είδους η κλίδα κατανομής εστιάζεται σε αυτές τις χειροπιαστές επενδύσεις. Με δεδομένες τις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και τα σχήματα της ε, αλλαγής τα τελευταία χρόνια έχουμε μια στροφή προς περισσότερα τέτοια, ε, προς, λιγότερο χειροπιαστές επενδύσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ταιριάζει σε αυτές τις αλλαγές η πρόταση και λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές και την ψηφιακή οικονομία. Βέβαια και αυτό που τελεί πρόκληση, πρόβλημα για την Επιτροπή για το τι δεδομένα μπορεί να δει, τι μπορεί να έχει για αυτού του είδους τις ε, χειρόπιαστες ή μη επενδύσεις. Να ένα αδύνατο σημείο. Άρα θα πρέπει ακριβώς να καλυφθούν και αυτές οι επενδύσεις από την κλίδα. Και επίσης να δούμε το πώς δεν θα τιμωρηθούν οι εταιρείες, δεν θα θυγούν οι εταιρείε όσον αφορά την περιουσία τους, το κεφάλαιό τους και έτσι να μην έχουμε Ιδίω τώρα που χρειάζεται αρνητικά, αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την ροή κεφαλαίων. Ακριβώς το χρόνο σας παραμείνατε. Μπράβο σας. Ο κύριος Χιούμερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να ξεκινήσουμε με τις βασικές σκέψεις. Όταν απευθυνθήκαμε στα μέλη μας να μας πούν ποιοι είναι οι βασικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά. Μίλησαμε για το ότι υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις στους 27 ή στους 28 όπως και για το ΦΠΑ και είναι προκειμένου. Έχουμε διαφορετική φορολογία και αυτό είναι τροχοπέδι για τις μη μη ε. Άρα το κόστος συμμόρφωσης είναι το πρόβλημα και όχι το φορολογικό βάρος. Από την αρχή επομένως ήταν επιθυμητό να υπάρχει μια ενοποιημένη κοινή βάση. Και εκεί τα πράγματα κόλλησαν στο Συμβούλιο. Άλλος λόγος τώρα που πάντα ήμασταν υπέρ αυτής της βάσης είναι όσα ακούσαμε από τον εισηγητή Τάγκ. Γιατί 27 διαφορετικά συστήματα σημαίνει ότι οι εταιρείε έχουν 27 δυνατότητες να έχουν τέτοιο φρολικό προγραμματισμό που θέλουν. Και άρα θα υπάρχει υψημένο κόστος συμμόρφωσης. Γι' αυτό και είχαμε επικριτική στάση για την πρώτη πρόταση της Επιτροπής. Εκεί που υπήρχε διακριτική ευχέρεια της χρήσης αυτής της κοινής βάσεις, το 11 αυτά. Όμως τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Και άρα για μας αυτό είναι πολύ θετικό ότι τώρα είναι υποχρεωτική αυτή η ρυθμίση για τις μεγάλες εταιρείε. Και οι ΜΜΕ έχουν ακόμα την κριτική ευκαιρία. Που μένουν σύνολο στις εθνικές αγορές, οπότε ίσως διέπονται από διαφορετική κατάσταση. Όμως θα πρέπει τώρα να μην ξεχνούμε το εξής. κάποια κρατημέλη δεν θα θέλουν να έχουν παράλληλα συστήματα. Σε περίπτωση που εγκριθεί αυτή η πρόταση, θα έχουμε κάποια κρατημέλη τα οποία δεν θα θέλουν να έχουν παράλληλα και την διακριτική, την, την προαιρετική ρύθμιση για τις ΜΜΕ. Δεν θα θέλουν δύο συστήματα και το σύστημα δεν θα πρέπει να γίνει υπερβολικά περίπλοκο γιατί θα πρέπει τα ΜΜΕ να μπορούν να συμμορφωθούν. Όχι, δεν θέλουμε να καλύφθουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό το καινούριο μοντέλο θα πρέπει να καλύψει και τις μικρότερες επιχειρήσεις. Και στις χώρες που δεν θέλουν δύο διαφορετικά συστήματα. Άλλο, οι ΜΜΕ θα ήθελαν, όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις, να ισχύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η κοινή βάση. Βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα Τέλο πάντων, αν αυτό είναι το καλύτερο που θα καταφέρουμε, για να αυτό είναι ο μόνο τρόπο να καταφέρουμε το σκοπό μα, τότε να δεχτούμε για κάποιο διάστημα το να μην ισχύει η ενωπημένη βάση, η κοινή βάση. Και αν επιτρέπεται κάποιο είδου αντιστάθμιση για τι διασυνορικέ απώλειε. Και βέβαια, καλύτερα είναι και δύο οδηγίε με μια να εγκριθούν. Επίσης, την ενιαία ρύθμιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση χρέους αλλά και το κεφάλαιο, το ενεργητικό των εταιριών. Οπότε και εδώ μας βγουν συμφωνούς οι προτάσεις της Κομισιόν από την άλλη μεριά. έχουν επιφυλάξει κάποια μέλη του φορέα μας όσον αφορά την τρέχουσα πρόταση. Όσον αφορά το τι εκπίπτει από τα κόστη ή τις δαπάνες έρευνας κλπ. Γιατί είπαμε ότι με την έκπτωση των δαπανών βοηθά έρευνα και ανάπτυξη. Και αυτό θα ωφελήσει κάποιες εταιρείες ε, οι οποίες έτσι αποκομίζουν κέρδη. Αλλά για τις νεοφυείς, startups, για διάφορες μικρές επιχειρήσεις αυτό δεν είναι καλύτερη ιδέα. Εκεί που υπάρχουν ε, κάποια project ε, και, καινοτόμα. Δεν έχουν αυτές οι εταιρείε κέρδη τη σχετική περίοδο. Άρα αυτή η ρύθμιση δεν είναι τόσο εύστοχη για αυτές τις εταιρείε. Δεν είναι πιο δόκιμη προσέγγιση. Ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω το θέμα, μήπως και το αλλάξουμε τώρα. Οι προτάσεις Λαμασούρ όσον αφορά ε, τις μη χειροπιαστές επενδύσεις, τις άειλες τέλος πάντων, και το αν μπορεί να ε, ε, εξασφαλιστεί ευελιξία μέσω των ε, νομοθετημάτων αυτών, των οδηγιών. Δηλαδή, συμφωνώ με τον προελέστατο συνάδελφο. Ευχαριστώ. Κύριε Χίμερ, ευχαριστούμε. Ο επόμενος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συμβάλλουμε στο έργο σα για τη βελτίωση τη φορολογική πολιτική στην Ευρώπη. Έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα ε, προσιλωμένη η οργάνωση την οποία εκπροσωπώ. Θα ήθελα για να κερδίσουμε χρόνο απλώς να σημειώσω ότι οι μέλη μας είναι όχι μεμονωμένοι φοροτεχνικοί λογιστές, αλλά ε, φορείς, οργανώσεις που εργάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ λοιπόν στο CCCTB στις ε, στις ε, ε, ενοποιημένες βάσεις. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε χαμένους και κερδισμένους στην αρχή. Η δια... επιλογή μεταξύ βραχυπρόθεσμης δυσκολίες και μακροπρόθεσμου συλλογικού κέρδους βέβαια δεν είναι δίλημα το οποίο έχει μπορέσει μέχρι τώρα να λύσει ικανοποιητικά η Ήπειρος και έτσι θα πρέπει να εξετάσουμε και πώς το CCTB θα καταστεί ε, αποδεκτό σύστημα για τα κράτη-μέλη εκείνα των οποίων η φορολογική ανταγωνιστικότητα αποτελεί λίδη αλήθεια της οικονομίας τους. Ε, είναι απλές, ευανάγνωστες οι προτάσεις. Για φορολογικό δίκαιο είναι κάτι το ασύνηθες αλλά πολύ ευπρόσδεκτο. Έτσι λοιπόν μια γραμμή πίστοσης έρευνας και τεχνολογίας για τις μικρές ε, νεοφυής. Είναι μια καλή προσέγγιση, αν και θα χρειαζόταν μια αξιολόγηση συνεπειών ή μια αντίστοιχη μελέτη. Πάντως πρέπει να διορθωθεί η μεροληπτική στάση απέναντι στο χρέος και τα χρεόγραφα και νομίζω ότι δεν πρέπει το κόστος να καταστεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάλογα υψηλό. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μπορούν να αποδειχθούν ε, στοιχεία τα οποία θα καταστήσουν το CTB πάρα πολύ χρήσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και πολύ θέλουμε βεβαίως να υποστηρίξουμε. Πέραν αυτό θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα χαιρετίζουμε την ε, πρωτοπορία που δείχνει και η Επιτροπή και οι Επιτροπέ ΕΚΟΝ και ΤΑΞΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται διεθνή συνεργασία, διαφάνεια και ευφυή ε, νομοθετικό σχεδιασμό. Η διεθνή συνεργασία καταρχά, η αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της φοροαποφυγής ε, ιδιαίτερα εξαρτάται από μια αναστονισμένο τρόπο προσέγγιση σε διεθνέ επίπεδο και ιδιαίτερα εδώ καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της ομάδας ε, κώδικα συμπεριφοράς. Επίσης η ιδέα της Επιτροπής Τάξη για τη θέσπιση ενός κέντρου συνοχής της φορολογικής πολιτικής και συντονισμού αυτής θα ήταν πολύ χρήσιμη. Ταυτόχρονα χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, για να αναφερθώ και στο δεύτερο κεφάλαιο, καλύτερη διαφάνεια σε όρου φορολογικού. Θα θέλαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τι σχετικές προτάσει για μια δημόσια αρχή, αλλά και να υποστηρίξουμε τι εταιρείε εκείνε οι οποίε έχουν εθελοντικά δημοσιεύσει εκθέσει αναχώρα. Εκείνοι οι οποίοι προάγουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό θα πρέπει να αποκαλύπτουν, να δημοσιοποιούν αυτά τα σχέδια. Πέραν αυτού όμως έχουν και οι ίδιοι την υπευθυνότητα, την ευθύνη για τα φορολογικά τους, αφού μόνο αυτοί γνωρίζουν ποιοι είναι οι, ποιες είναι οι πραγματικές λεπτομέρειες της υπόθεσης του φορολογικού σχεδιασμού. Ε, μια εφίς λοιπόν νομοθεσία ως τρίτο κεφάλαιο που θα πρέπει να ε, υπαγορευθεί και να υποστηριχθεί και με κυρώσεις. Θεωρώ ότι ένας κώδικας συμπεριφορά μπορεί να και πρέπει να καλύπτει και τις ε, υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, αλλά θα πρέπει να καλύπτει όλους τους παρέχοντες τέτοιε υπηρεσίες με βάση και τη δραστηριότητα, όχι μόνο τον τίτλο μιας ε, επαγγελματική κατηγορίας ή τομέα. Ιδάλλως δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος του δημοσίου συμφέροντος. Ε, Επίση οι κανόνες που αφορούν την εξασφάλιση για τις φορολογικές αρχές ε, υποστήριξης από τις υπηρεσίες ε, δημοσιονομικού ελέγχου είναι πολύ περιοριστική σε σχέση με το νέο κανονισμό 537-2014 και χρειάζεται να ενισχυθούν περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω κλείνοντας ότι οι επαγγελματίες λογιστές ιδιαίτερα σοβαρά βλέπουν το ρόλο τους και τις ευθύνες τους στο, στην καθημερινή μας πρακτική. Η μεγάλη πλειονότητα των επαγγελματίων λογιστών δρά κατά τρόπο καθοριστικό για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων παρά την ε, περιπλοκότητα τους ε, εξασφαλίζουν να μπορούν οι φορολογούμενοι να πληρούν τις ε, υποχρεώσεις τους και θεωρούμε ότι μια αποτελεσματική χρήση πόρων αλλά και τήρηση δεντολογικών προδιαγραφών είναι δεδομένη. Ως επαγγελματική τάξη λοιπόν είμαστε ε, προσιλωμένοι στο δημόσιο συμφέρον και είμαστε στη θέση σας για οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους με τα σχόλιά τους. <laughs> Λυπούμε, αλλά ο πρώτος είμαι εγώ. Και θα μιλήσω γερμανικά τη μητρική μου γλώσσα. Έχω κάποια θέματα στα οποία θέλω να τοποθετηθώ. Ε, συμβολή στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ε, χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια ή από δαπά κεφάλαια. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διάκριση και δεύτερον μήπως είναι προκυκλικό το στοιχείο αυτό. Μήπως τελικά δηλαδή πιο πολύ ζημιά κάνουμε παρακαλώ. Επίσης η άνηση αντιμετώπιση της χρηματοδότησης από όλο από πόρους αντί για ιδίους πόρους γιατί πρέπει να μπει σε μειονεκτική θέση. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει νόημα να μπουν σε αυτό το ε, σύστημα με την υποχρέωση λογοδοσίας που μπορεί να είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. Φερρυπίν, το γερμανικό, ο γερμανικός εμπορικός κώδικας ε, μπορεί να έχει τελείως διαφορετικές θέσεις και προτάσεις ή όρους από άλλες νομοθεσίες. Η ενοποίηση <coughs> επίσης ε, είναι χρήσιμη και πάλι αυτό σε αντιπαράθεση με τον γερμανικό εμπορικό κώδικα. Τα άειλα, αγαθά, άειλο ενεργητικό δεν ε, περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής και αυτό γίνεται σκεμμένα. Πλην όμως στην ε, τωρινή μορφή της οικονομίας, ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις, έχει πολύ μεγάλη, αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία το άϊλο ενεργητικό, ε, ευρεσιτεχνίας ε, κλπ. Μπορούμε να τα γνωρίσουμε λοιπόν αυτά ή μήπω πρέπει να καλυφθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Προς τον τρίτο εκπρόσωπο κυρίως των, ε, του Accountants Europe απευθύνεται αυτή η ερώτηση. Αυτέ ήταν οι δικέ μου λοιπόν ερωτήσει. Θα ακούσουμε και του συναδέλφου και θα σα δώσω το λόγο στο τέλο των ερωτήσεων για να απαντήσετε. Και τώρα ξαναγυρνάω στα αγγλικά. Ελπίζω να τήρησα τον δικό μου χρόνο που ήταν δύο λεπτά να ομιλητή. Ελπίζω να μην, να μην μίλησα πολύ γρήγορα για του διερμηνεί. όχι. Και προχωρώ στον Νίκ Μπαγιέ από του Ελληνιστές Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου όσου πήραν το λόγο για τι εξηγήσει που έδωσαν. Είναι σημαντικό θέμα που επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα είναι σημαντικό να ακούσουμε του διάφορου φορεί που άμεσα εμπλέκονται. Ακόμα και ότι στον τομέα σα είναι δύσκολο να υπάρχει μια ομόφωνη θέση, αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε διάφορου τρόπου, ώστε να καταλήξουμε σε καλύτερη φορολογική δικαιοσύνη, συνεχίζοντα να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Όταν είμαστε δημοκράτε, όπω είμαστε εμεί, η πολιτική δεξιά και αριστερά, σε δύσκολε στιγμέ, περνάμε δύσκολε στιγμέ να προσπαθούμε να εξηγούμε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει που είναι το 85-90% τη οικονομία στην Ευρώπη Πώ γίνεται να πληρώνουν 30% παραπάνω φόρου από ό,τι οι πολυεθνικέ. Άκουσα κυρίω τον εκπρόσωπο τη Business Europe, άκουσα αυτά που μα είπαν, με τα χαρά άκουσα το ότι υπερσπεζόσαστε την ενοποίηση, το τι μα ενοποίησε, συμφωνώ μαζί σα, πιστεύω ότι αυτό θα μα επιτρέψει να πλησιάσουμε καλύτερα τα διάφορα προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη ευρωπαϊκή οικονομία, που είναι το φορολογικό σύστημα που δημιουργεί πρόβλημα στο κείμενο της ενοποίησης ε, για την ώρα δεν υπάρχει κοινό ποσοστό για, κάθε, για όλες τις χώρες. Κάθε χώρα καθορίζει το ποσοστό φορολόγησης. Μήπως ε, θα ήταν πιο σωστό, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, να υπάρχει ομοσπονδιακό, ε, ομοσπονδιακός φόρος που θα είναι ίδιος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με μια διαμόρφωση ανακάτω μέλος 5 με 10% ούτως ώστε να γίνει ένα πρώτο βήμα και έτσι όλοι θα αντιμετωπίζονται ισότιμα. Το δεύτερο ερώτημα, πιο γενικό και απευθύνεται ίσως πιο ιδιαίτερα προς την Business Europe, είναι το εξής. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ τζίρο είναι υποχρεωτική αυτή η φορολόγηση. Είναι κάπως παράξενο, διότι υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, κέρδος κάτω από 750 εκατομμύρια ευρώ αλλά που έχουν διεθνείς δραστηριότητες και δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες. Ε, θα ήθελα να ξέρω λοιπόν κατά την άποψή σας μπορούμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτό το όριο για να έχουμε μια φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη. Τελευταία ερώτηση κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος. τον κύριο Μνέρ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι σκέφτονται για αυτό το κείμενο, διότι τις αφορά μέσα και θέλουμε να τις βάλουμε σε ίση βάση όσον αφορά τη φορολόγηση με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να προσέχω το χρόνο, λέει ο Πρόεδρος, διότι έχουμε μια κοινή συνεδρίαση μετά και δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε. Επόμενος, Σάντερ Λούντς για το ECR, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω τον θεμητό φορολογικό ανταγωνισμό, μειώνεται έτσι ο φόρος και τα κράτη-μέλη προσπαθούν να είναι πρώτα και ανταγωνίζονται. Αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις μετά αυτά που άκουσα ο χρόνος αγόρας είναι περιορισμένος, ακούσαμε περισσότερο γενικές δηλώσεις. Θα ήθελα να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι άκουσα πολλές ε, ισχυρές δηλώσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε ότι το σύστημα θα δώσει ασφάλεια δικαίου και ένα σύστημα ασφάλες και δίκαιο ε, και θα έχουμε νομική ασφάλεια δικαίου. Πώς μπορούμε να λύσουμε, να πούμε ότι θα έχουμε ένα σύστημα μάλλον που είναι δικαιότερο. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να γίνει και προς τον κύριο Βάτσον είπατε ότι ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη θα χάσουν. Διαβάζοντας το έγγραφο τοποθέτησης βλέπω ότι εκεί αναφέρεστε σε απόλυτη ευελιξία τα κράτη-μέλη, κυρίως για τα μικρότερα κράτη-μέλη. Άρα θα ήταν ενδιαφέρον ε, να γνωρίζουμε γιατί οι επιχειρήσεις των μικροτέρων κρατών μελών θα πρέπει να φοβούνται ότι θα χάσουν περισσότερα μιλάμε για οικονομική σύγκληση στο Κοινοβούλιο πολύ. Το συζητούμε διαρκώς και δεν θα έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση αν μετακινήσουμε επιχειρήσει από τα μικρότερα κράτη-μέλη προς τα μεγάλα κράτη-μέλη που είναι ήδη ισχυρά οικονομικά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μετά έγιναν κάποιε δηλώσει για το διοικητικό κόστο και το διοικητικό άχθο. Τα ανέφερε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι, όπω ο κύριο Μπουτέλη Ταφτ, όπου είπε ότι θα έχουμε ένα σύστημα που είναι απλούστερο, σαφέστερο και έχουμε την εξαιρετική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Φαντάζομαι ότι στο νέο σύστημα οι πολυεθνικές, παρά το ότι έχουν το CCCTB, θα είναι υποχρεωμένες να προετοιμάζουν και ε, εγχώρια λογιστικά και να υποβάλουν δηλώσεις σε επίπεδο κράτους μέλους. Πώς θα είναι αυτό απλούστερο και δεν είναι πρόσθετο διοικητικό άκθος, το καταλαβαίνω επ' αυτού. Αν ο κ. Μπουτέλη Ταύτη είχε την καλοσύνη να πει περισσότερε λεπτομέρειε, θα με ενδιαφέρε να τι ακούσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο, Λίβε Βίρινγκ για του ε, φιλελεύθερου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, όταν μιλάμε για τη φορολόγηση πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πιο δίκιο ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών η καλύτερη λύση εδώ θα ήταν να συνδέσουμε τη φορολόγηση επιχειρήσεων με την οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκολύνουμε τις εταιρείε να μπορούν να επιχειρούν, να κινούνται εντό τη εσωτερική αγοράς. Οι διεθνείς εταιρείε χρειάζονται έναν αρμονισμένο σύστημα με κοινού ε, κανόνε. Η διάβρωση της φορολογικής βάσεως είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμηθεί. Όλοι πρέπει να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιο του όσον αφορά του φόρου και εταιρείε. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή την πρόταση για το CCCTB. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο φόρο των επιχειρήσεων είναι σημαντικό για τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και είναι ένα έσοδο πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ένα ιδεώδη σύστημα που ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Έχω κάποιες ερωτήσεις στον φάτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, πόσο σίγουρη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόταση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, ότι δεν θα έχει καμία επίπτωση όσον αφορά την κατάσταση που κρατεί στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη και τα παρόντα και τα μελλοντικά ενδεχόμενα για τα κράτη-μέλη, καθώς και το περιθώριο ελιγμών που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, ε, υιοθετώντα μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι δημοσιονομικά οδέτερο. Δεύτερον, θα ήθελα να γνωρίζω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη την ψηφιακή οικονομία ε, παρουσιάζοντας αυτές τις προτάσεις. Οι προτάσεις τις λαμβάνουν υπόψη εταιρείε που χρησιμοποιούν ρομπότ οι εταιρείε οι οποίε πολλούν ευρωπαϊκά big data ή λογισμικό λαμβάνει υπόψη τα πνευματικά δικαιώματα και πώς η οικονομική αξία αυτών εκτιμάται και πώς αυτό μεταφράζεται στα μέτρα που προτείνονται. Και τελική ερώτηση. Οι εταιρείε θα συνεχίζουν να προσπαθούν να βελτιστοποιούν το καθεστώς το φορολογικό τους. Να μην είμαστε αφελείς με το CCCTB θα το κάνουν αυτό μέσω των μέτρων και το, της ε, φορολόγησης εταιριών θα πηγαίνουν να εγκαθίστανται στις χώρες εκείνες που έχουν το χαμηλότερο φόρο των επιχειρήσεων. Οπότε θα οδηγήσει σε μια κάτωθη κίνηση. Το λέω αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Μετ Καρθή. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τους ομιλητές για το όσα μας παρουσίασαν και όπως άλλοι προλαλήσαντες και εμείς προβληματιζόμαστε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του CCTB σε σχέση με το κατά πόσο θα καταπονήσει την ε, φοροδιαφυγή ε, και ιδίω αυτά τα 750 εκατομμύρια και επίσης κατά πόσο πρόκειται αυτό να βοηθήσει ε, στις επενδύσεις και τι θα γίνει και με τις δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης, πάρα πολλοί στην Ιρλανδία έχουν επιφυλάξει αυτή την πρόταση και για τις επιπτώσεις που θα έχει στο εισόδημα σαν αποτέλεσμα του, δικού μας ε, στραβλού μοντέλου. Ε, να υπάρξει αλλαγή και η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα από το CCTB είναι δύσκολο να υπολογιστούν όσον αφορά την Ιρλανδία αλλά και άλλες χώρες. Ε, άκουσα τις ε, απόψεις των ομιλητών και έχουμε αυτές τις εκτιμήσεις για το εισόδημα της Κομισιόν αλλά δεν είναι τόσο αξιόπιστα όσον αφορά τα fixed tangible assets, αυτά τα χειροπιαστά ε, στοιχεία ενεργητικού, ε, ιδίως όσον αφορά την βιομηχανία, τι θα γίνει με την αεροναυπήγηση επίσης. Και όσον αφορά το άρθρο 40 και αυτό το 10% της αξίας των χρηματοπιστωτικών ε, περιουσιών και στοιχείων ενεργητικού είναι δυνατόν αυτές οι επενδύσεις να μετατραπούν σε τέτοια στοιχεία. Πέστε μας τι ισχύει. Μήπως έχετε κάποια άποψη για το τι μπορεί να γίνει ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανασχέσουμε τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις Σβενγκίγκολτ για τους πρασίνους. Η Εύα, η Εύα Ζολή. Η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τον εκπρόσωπο του Business Europe, κύριο Γούτσον. Είστε υπέρ του να γίνει μια τέτοια μεταρρύθμιση, ναι, αλλά προτιμάτε το σύστημα να είναι προαιρετικό, ούτως ώστε κάθε επιχείρηση να διαλέξει τι τη συμφέρει, το εθνικό σύστημα ή το σύστημα CCTV. να μην γίνουν όμως τα πράγματα πιο περίπλοκα, να μην αυξηθεί ο διοικητικό λαβύρινθος, αφού αυτό που θέλουμε είναι τη μείωσή του και θέλουμε να είναι φεμιτές οι συνθήκες του ανταγωνισμού. Για το, το, το, τον εκπρόσωπο του ΕΜΠΕ, το 2011 ήσασταν υπέρ της πρώτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το ότι ήταν πολύ περίπλοκη όσον αφορά την εφαρμογή τη για τις ΜΜΕ. Ισχύει αυτό ακόμη κατά την γνώμη σα. Αυτή η πρόταση του 2016. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα στις ΜΜΕ ε που δρούν σε πάνω από μία χώρα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα προσκεκλημένοι μας μπορούν να απαντήσουν όλες αυτές τις ερωτήσεις με την ίδια σειρά να το κάνουμε. Οπότε παρακαλώ απαντήστε στα πιο βασικά, μια που ήδη είμαστε ελαφρώ πίσω στον πρώτο χρονοδιάγραμμα μα, κύριε Βότσον. Ξεκινούμε με την ερώτηση των Πρασίνων. Είναι αλήθεια, όταν είχαμε την προηγούμενη πρόταση, λέγαμε ότι θέλουμε να συνεχίσει να είναι προαιρετικό. Έχουμε τώρα τι θέση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λέμε ότι υπάρχει πρόταση να είναι προαιρετική ρυθμίση για όλου. Αλλά αυτό να μην είναι προπόθεση. Όχι. Αλλιώς θα φτάσουμε να πούμε όχι στην πρόταση. Να μην υπάρχει τέτοιου είδους διπλή ρυθμίση για όλους. Έτσι αντιλαμβανόμαστε αυτό το έγγραφο της Κομισιόν τώρα. Όσον αφορά τα άειλα της επενδύση, αυτό που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτά τα εκάλυψα στην ε, παρουσίασή μου. Επίσης ε, πολλά ακούγονται για κερδισμένους και χαμένους. Εγώ θα σας έλεγα, κοιτάξτε, που κατέληξε το κοινό κέντρο ερευνών της Κομισιόν. Νομίζω ότι εκεί έχουμε στοιχεία ε, σημαντικά για κερδισμένους και χαμένους. Νομίζω ότι μπορούν οι συνεργάτες σας να σας ε, παρουσιάσουν αυτή τη μελέτη. Τώρα άλλο. Από τα μπροστινά έδρανα πάντοτε με εκπλήσει όταν ακούω τέτοιε διατυπώσει όπω α πούμε το ότι τα φυσικά πρόσωπα πληρώνουν περισσότερο από ότι οι εταιρείε. Για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά λίγο πιο αποστασιωμένα. Ποιοι είναι οι κύριοι αυτών των ε, εταιριών. Άνθρωποι είναι. Πολλές φορές μιλάμε για τα κέρδη των εταιριών. Ε, αυτά τα κέρδη είναι φορές για τις συντάξεις των εργαζομένων. Τίποτα δεν δίνεται τζάμπα. Άρα, άμα αυξήσουμε τον εταιρικό φόρο, θα πληρώσουν την ύφη τα φυσικά πρόσωπα. Οπότε, για να σκεφτούμε τι σύστημα εταιρικού φόρου ισχύει και πώς αυτό επιδρά το γενικότερο σύστημα. Ναι, στις τη εταιρείε είναι χαμηλότερος από ό,τι για τα φυσικά πρόσωπα. Αλλά κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει μετοχές και πληρώνει δύο φορές. Γιατί πληρώνει και μέσω του εταιρικού φόρου. Και αν λειτουργεί σωστά ο φόρος τότε πληρώνει ξανά όταν παίρνει το μέρισμα από τα κέρδη αυτό το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Άρα να προσέχουμε να κάνουμε αυτέ τι διακρίσει όταν κρίνουμε τα συστήματα φορολόγηση φυσικών προσώπων και εταιρεών. Τώρα για τα κατόφλια. Όσον αφορά αυτέ τις ε, αναχώρα κοινοποίησεις. Να δούμε το θέμα γενικότερα. Το Business Europe είναι υπέρ της πρότασης της Κομισιόν όχι, συγγνώμη, κύριος ο ομιλητή την πρόταση του ΟΣΑ όσον αφορά τις κοινοποίησεις, τη δημοσιοποίηση αναχώρα. Και κάτω κάνει την πρόταση της Κομισιόν και νομίζω ότι οι φορολογικές αρχές είναι η σωστή ε, πλατφόρμα, η σωστή αρχή για να καταλήξουν αυτές οι πληροφορίε από τις εταιρείε. Και συμμορφώνονται οι εταιρείε με την φορολόγηση. και είναι συμφέρον των εταιριών να υπάρχουν θεμητοί όροι ανταγωνισμού. Αλλά ακόμα δεν έχουμε πιστεί ότι στέκει αυτού του είδους η δημόσια κοινοποίηση ανά χώρα. Μήπως και έτσι υπονομεύεται η δουλειά των φορολογικών αρχών, το καθημερινό του έργο. Είναι σαν λέει ότι δεν μπορούν να δουλέψουν οι φορολογικές αρχές εάν δεν υπάρχει εποπτεία. σε αυτές τις πληροφορίες. Μα έτσι δύσκολα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου το φορολογικό σύστημα ή τέλο πάντων οι φορολογικές αρχές. Με αυτό κατά νου θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ρύθμιση αυτής της κοινοποίησης. Ξέρετε, ασχολούνται δύο επιτροπές με αυτό και θα πρέπει να δούμε το πώς αυτού του είδους η δημόσια κοινοποίηση θα προχωρήσει και να δούμε τα κατόφλια θα βοηθήσουν ε, στην διαφάνεια και τώρα ξέρω ότι κυκλοφορεί αυτή η πρόταση ότι όταν κατέβει ακόμη αυτό το όριο, αυτό το κατόφλια ε, θα βοηθήσει αλλά προσοχή γιατί ελοχεύουν κίνδυνοι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις ε, διευκρινήσεις σας ο κύριος Χιούμελ. Μια και έχω και ένα λεπτό παραπάνω από το Μάικ, θα απαντήσω σύντομα σε ερωτήσει. Πρώτον, για την ομάδα των Πρασίνων και τοποθέτησή τη. Εμεί, όσοι ΑΠΜΕ, έχουμε επικρίνει την πρόταση κυρίω λόγω τη ε, εθελοντική πλούσιας ευκαιρίας που δίνει για συμμετοχή σε μεγάλε επιχειρήσει. Εκεί είναι το θέμα μα. Είμαστε υπέρ του, της υποχρεωτικής υπαγωγής και όχι της ε, δευτερον Δεύτερον, μικρά κράτη-μέλη. Πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση. Εάν έχει αρνητικές συνέπειες για ορισμένα μικρά κράτη-μέλη αυτή η πρόταση, αυτά τα οποία τώρα τεχνητά ε, ελκύουν, προσελκύουν επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις λόγω χαμηλού χαμηλής φορολογικής δάσης και τρίτον, εάν η Ιρλανδία έχουν τέτοιο κέρδος οι χώρες αυτές αλλά με την αλλαγή θα υποφέρει μόνο η χώρα, μόνο η Ιρλανδία εάν ε, αλλάξει η φορολογική βάση και δεν θα έχει πρόβλημα η επιχείρηση. Ε, ο Υπουργό Οικονομικών τη Ιρλανδία θα υποστεί τη ζημιά που θα, θα εισπράξει λιγότερα έσοδα για τη χώρα και όχι η επιχείρηση. Και για μένα μεγάλη σημασία έχει αυτό που ρώτησε ο ε, πρόεδρο για τις καινοτόμε μικρομεσαίες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και νομίζω ότι και άλλοι τηρούν προς αυτό το συμπέρασμα το εάν θα πρέπει να αλλάξουν οι λογιστικοί κανόνες με την υπαγωγή. Να το πω αλλιώς. Εάν θέλει μία μικρομεσαία επιχείρηση να αναπτύξει διεθνείς δραστηριότητες και άρα να προσελκύσει τις κεφαλαϊκές αγορές. Καλό θα ήταν να αρχίσει να σκέφτεται να αλλάξει τους κανόνες, τους εταιρικούς στο EFAS και να μπει στο σύστημα αυτό, να υπαρθεί στο σύστημα. Εάν θέλει να μείνει στο εθνικό μόνο επίπεδο με μικρές διασυνοριακές συναλλαγές μόνο, δεν την ε, συμφέρει να μπει στο διεθνές σύστημα. Το ε, ερώτημα όμως τι θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση σε χώρες, όχι όπως η Γερμανία, Φερρυπίνα, αλλά να, η Γαλλία, η Αυστρία και άλλες χώρες επισημαίνουν ότι δεν είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν με δύο παράλληλα συστήματα λογιστικά στο μέλλον γιατί θα είναι διαφορετικές οι βάσεις, διαφορετικές και τα διαφορετικές και νομοθετικές βάσεις, αλλά και οι φορολογικέ βάσεις και είναι δύσκολα διαχειρίσιμο ένα τέτοιο σύστημα για το μέλλον. Άρα οτιδήποτε συζητούμε τώρα για το περιεχόμενο του συστήματος αυτού θα πρέπει να το δούμε και με προβολή στο μέλλον, ε, εάν είναι δυνατόν να ε, εφαρμόζεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όπως είπαμε, πολλές ε, χώρες σκοπεύουν να εφαρμόσουν το ίδιο σύστημα σε όλες τις εταιρικέ μορφές, ακόμα και τις πολύ μικρές. Και επίσης για τον εκπρόσωπο της ομάδας των φιλελευθέρων. Θα ήθελα να εκφράσω προτίμηση στο να μετακινείται κάποιος προς χώρα όπου είναι χαμηλότερος ο φόρος στη φάση την τωρινή όπου μπορεί να έχει περισσότερο κέρδος γιατί έτσι είναι πιο διαφανής ο ανταγωνισμός μεταξύ των όρων. Και άρα και τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται σε μια αποτελεσματική και υπεύθυνη ε, χρήση των ε, χρημάτων που πληρώνει ο φορολογουμενός τους. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν διατυπώσει πολλές ε, και σημαντικές ερωτήσεις. Δεν μπορέσω να τις ε, εξαντλήσω όλες. Αν μου επιτρέπετε όμως, θα επικεντρωθώ σε αυτές που θεωρώ πιο σημαντικές. Το διοικητικό βάρος, το διοικητικό κόστος ε, που πολύ σωστά επισήμαναν αρκετοί ομιλητέ. πρέπει να το κοιτάξουμε. Η πραγματικότητα των εταιριών είναι αφενός μεν ότι θα πρέπει να προετοιμάζουν γενικές οικονομικές ε, ή φορολογικές καλύτερα και σε άλλες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν σχετικές προσαρμογές για να ανοίξουν τη φορολογική βάση. Μόνο στις ε, λεγόμενες συγμένες ε, εταιρείε της Ευρώπης έχει εξασφαλιστεί συμφωνία για τα διεθνή πρότυπα, συλλογικά θα έλεγα. Και εδώ η Ευρώπη έχει πρωτοπορία επιβάλλοντας την εφαρμογή των παγκόσμιων προδιαγραφών. Αυτό μπορεί να μας βάλει σε σκέψεις, γιατί όταν φτάσουμε στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες δεν εφαρμόζουν το διεθνές σύστημα και πρέπει να συζητήσουμε την οδηγία για τα λογιστικά πρότυπα, τότε και εδώ και στο Συμβούλιο νομίζω δεν θα μπορέσετε να καταλήξετε συμφωνία. Το αποτέλεσμα ήταν μια οδηγία με πάνω από 100 διαφορετικές επιλογές που απεδεικνύει έτσι πόσο διχασμένα ήταν τα κράτη-μέλη μεταξύ του και έτσι άφηνε και ένα πολύ ευρύ περιθώριο προσαρμογή διακριτική ευχέρεια μεταξύ των κρατών μελών. Καλό λοιπόν θα ήταν να έχουμε μεγαλύτερη πρόοδο με μια έμεση συνέπεια την ευχερέστερη φορολογική προσαρμογή. Ταυτόχρονα σημαντικό ερώτημα ήταν αυτό το οποίο φορούσε το άειλο ενεργητικό που θα πάρει πολύ μεγαλύτερη σημασία πιστεύω στο μέλλον από ό,τι μέχρι τώρα και εδώ χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά όχι μόνο για το πώς θα αναγνωρίζετε το άϊλο αυτό, πώς θα καταγράφετε το άϊλο αυτό ενεργητικό, αλλά και πώς θα υπολογίζονται οι μεταβιβάσεις, γιατί μην ξεχνάμε είναι το πιο, ευ... το πιο ε, πτυτικό ή κινητικό, αυτό που πιο εύκολα μεταβιβάζεται. Και εδώ χρειάζεται πιστό συντονισμό σε διεθνέ επίπεδο. Στην ε, διαχείριση, στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζετε αυτό από την νομοθεσία. Επίσης, εν ώψη και της ε, συζήτησης για τις φορολογικές αρχές, πρέπει να πω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα όχι μόνο στατικά, αλλά να κοιτάξουμε και τις μελλοντικέ γενιές. Θα ήταν ε, λυπηρό λοιπόν ένα σύγχρονο ε, φορολογικό σύστημα να μην κοιτάξει και τι προσθέμενη αξία προσφέρουν οι επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές, περιβαλλοντικό αντίκτυπο, παραδείγματι, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη μετάβαση προς μια πιο αηφόρο οικονομία. Για τους ε, κερδισμένους και τους χαμένους που ακούστηκαν πολλές φορές, αναφέρθηκαν, το θέμα δεν είναι να κρατήσουν περισσότερο οι συζητήσεις. Το θέμα είναι να συζητήσουμε μια μεταβατική περίοδο, ώστε κράτη τα οποία περισσότερο έχουν βασίσει την οικονομία τους σε μια φορολογική ανταγωνιστικότητα, σε ένα φορολογικό να έχουν το περιθώριο να προσαρμοστούν. Λοιπόν, πάρα πολλέ διαδικασίε πολιτικέ θα ξεκινήσουν. Φτάνουμε στη δεύτερο μέρο, Κάτια Λεχτοκόμουνάινεν από την ΕΤΟ και Ρίτσαρτ Μέρφυ, μέλος του Tax Justice Network. Ένα πεντάλεπτο ανακεφάλι για μια εισαγωγή και μετά θα ακολουθήσουν οι ομάδες. Κάτι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Δύο βασικοί τομείς είναι αυτοί που καλύπτουν τις φωτές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενδιαφέρονται πολύ τα μέλη των συνδικάτων. Για το φορολογικό τομέα ενδιαφέρονται και το κοινωνικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έχει κλονιστεί όπως λόγω του Brexit. Οπότε πρέπει όλοι να εργαστούμε την ένωσή μας. Και να δείξουμε ότι δεν αφορά μόνο την οικονομία προσπάθεια, αλλά και ισχυρά κοινωνικά δικαιώματα και πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν πράγματι τα προβλήματα φοροδιαφυγής. Τα μέλη του Συνδικάτου α, πρέπει να πληρώνουν α, φόρους. Είδαν ότι έχουμε περικοπές όμως στις δημόσιες δαπάνες και περικοπές στους μισθούς. Εξακολουθούν όμως τα μέλη μας να πληρώνουν τους φόρους. Άρα δίκαιον να μπορούν να βλέπουν ότι και οι πολυεθνικές πληρώνουν α, ε, τους ε, δίκαιους φόρους που τους ε, αρμόζουν, που τους, τους ταιριάζουν. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνη. Για να έχουμε αυτά αποτελέσματα, για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και το φορολογικό dumping και επιλογή φορολογικού θεστώτο, είναι ένα τρόπο να ξαναποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του λαού και πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω τρία βασικά σημεία να τονίσω. Πρώτο, στηρίζουμε εν γέννη το CCCTB. Δεύτερον, οι τροπολογίε μας όσον αφορά το CCCTB θα υποβληθούν και ε, ζητάμε να υπάρχει ένα κοινό φόρος για τις εταιρείε. Το ETUC στηρίζει ως προτάσεις που έχουν σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του φορολογικού dumping και επιλογή φορολογικού καταστώτο. Υποστηρίζει το ETUC, το CCCTB και την υποχρεωτική εφαρμογή αυτού. Προτείνουμε όμω και τροπολογίε. Οι αγορές από μόνες τους δεν οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα απαραίτητα. Αντιθέτως, ε, ε, έχουμε αρνητικά αποτελέσματα από το φορολογικό ντόμπινγκ φοροδιαφυγή. Το CCCTB είναι κάτι θετικό. Θεσπίζει κοινού κανόνες, όπως είπε και ο Μονταλία προηγουμένω για τις επιχειρήσεις ε, που κινούνται στην εσωτερική αγορά. Στο ETUC είμαστε υπέρ δίκαιων κανόνων και επιχειρήσεων που κινούνται βάσει των δίκαιων κανόνων τα μέλη του, τα συνδικάτα μας μπορούν να δείξουν ε, πόσο τεράστια είναι τα ποσά των απολυστέντων φόρων. Μπορώ αργότερα να αναφερθώ σε αυτά. Ο, ο καθηγητής Μέρφυ θα αναφερθεί σε αυτά. Έχουμε κάνει υπολογισμούς και είδαμε ότι οι φόροι που έχουν χαθεί αντιπροσωπεύουν 139,3% του συνολικού ελλείμματο του ετησίου τη Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αν είχαν συλλεχθεί αυτοί οι φόροι, δεν θα χρειαζόταν περικοπέ και οικονομικέ προσαρμογέ και θα μπορούσε να είχε συγκρατηθεί το, το έλλειμμα στον αφορά τα δημοσιονομικά. Οι τρει βασικέ μα τροποποίησεις που προτείνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το όριο, το κατόφλιο. Ζητούμε το όριο να καθοριστεί πολύ χαμηλότερα από αυτό που προτείνεται. Απαιτούμε και ζητούμε το κατόφλιο αυτό να καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες περιλογιστικών. Έτσι θα αυξηθεί η συνοχή και η σαφήνεια των κανόνων. Το κατόφλιο θα έπρεπε να είναι το πολύ στα 40 εκατομμύρια ευρώ. γεωγραφική κάλυψη. Ζητούμε η οδηγία να συμπληρωθεί για τις πολυεθνικές εταιρείες και στα κατί της Ευρωπαϊκής Ενώσης και σε τρίτες ε, χώρες και οι όμιλοι να καλύπτονται. Οι εταιρείε σε τρίτες χώρες που καλύπτονται ήδη από την οδηγία καταπολεμήσεως της φοροδιαφυγής αλλά όχι με έναν τρόπο τόσο φιλόδοξο όσο ζητούσε η TUC. Και κάτι άλλο αναφέρθηκε πριν. Σχέση μεταξύ του CCCTB και της υποβολής εκθέσεων αναχώρα. Το ETUC στηρίζει λεπτομερή υποβολή εκθέσεων αναχώρα με πλήρη διαφάνεια για όλες τις εταιρείε σε παγκόσμιο επίπεδο. Το CCCTP και εκθέσεις αναχώρα πρέπει να κινηθούν παράλληλα αποτελεσματικά για τη συλλογή επαρκών πληροφοριών που είναι πολύτιμες για κάθε χώρα συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών. Εταιρείε τι εννοώ εταιρείε που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Υποστηρίζουμε τι εκθέσει αναχώρα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ για διαφάνεια και για την καταπολέμηση τη μετακυλήσεω, μετακινήσεω των κερδών και τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ταχεία εφαρμογή. Ε, είναι μία από τι τροπολογίε που βάλαμε. Παροτρύνουμε γρήγορη εφαρμογή του CCCTP. Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή θα πρέπει να ξεκινήσει το αχύτερο δυνατόν από Ιανουάριο 2019. Μόνο με το CCCTB και την σωστή προσέγγιση θα αποφύγουμε τα προβλήματα. Υπάρχει το θέμα των λογιστικών, των κανόνων των λογιστικών. Ο κύριος καθηγητής το έχει ερευνήσει περισσότερο το θέμα αυτό. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό. Ζητούμε ένα, ένα κοινό ποσοστό φορολογής εταιριών. Εμείς ε, ζητούμε 25% περίπου. Τέλος. Κυρίες και κύριοι, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αξίζουν μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογήσεως ε, των ε, επιχειρήσεων και ένα κοινό ποσοστό φορολόγησης. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μέρφυ και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων για την έρευνα που έκανε για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. με το λόγο στον κύριο Μέρφυλε, ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε ως μέλος αυτού του δικτύου μας για την φορολογική δικαιοσύνη, αλλά και άλλες σήμερα ε, που παρίσταται σχετίζονται με μας Είμαι καθηγητής στο City University του Λονδίνου, οπότε ξέρετε ότι ήδη είμαι προκατηλημένος κατά αυτού του συστήματος, γιατί από την αρχή έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι θετικό το CCCTB. Το θέμα είναι ότι η σημερινότητα φόρο είναι σε έναν μύθο στριγμένο. Δηλαδή, οι όμιλοι εταιρεών αποτελούνται από ανεξαρτηστερίες, αλλά αυτό είναι ένα παραμύθι. Αυτό το παραμύθι πρέπει να το ξεχάσουμε και να σκεφτούμε ότι τελικά πρόκειται για ενιαίες οντότητες οικονομικές και υπάρχει κεντρική διαχείριση και θα πρέπει έτσι να φορολογηθούν. Άρα το CCCTV αναγνωρίζει ακριβώς μια οικονομική πραγματικότητα η οποία μέχρι τώρα απουσίαζε εδώ και δεκαετίες. Μόνο είναι αυτή τη ενία είναι αυτή τη που να προχωρήσουμε. Επίσης μην ξεχάσουμε το τι σημαίνει εταιρικό φόρος είναι ένας φόρος backstop. 8% του, των φορολογικών εσόδων ο λόγος που υπάρχει είναι για να μην υπάρχει ε, κάποιος φοροδιαφυγή σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος ο οποίος αλλιώς πρόκειται να έχει ε, δυναμητιστεί, να έχει <clears throat> σαμποδέστη. Οπότε ε, έχουμε τώρα κάποιους οι οποίοι κάνουν τις επιλογές τους και πάνε από κράτος σε κράτος και αυτό οδηγεί σε τεχνητό ανταγωνισμό. Για δούμε επομένως την πραγματικότητα. Ως οικονομολόγος να σας πω ότι τελικά οι εταιρείε χρειάζονται θεμητό ανταγωνισμό. Ιδάλλως έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό και σήμερα αυτό ισχύει γιατί δεν έχουμε συνεπή συνεκτική ρύθμιση. Το CCTB ε, άρα προ τα εκεί πάει, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι αυτό το τρίτο C, η ενοποίηση. Η πρόταση αυτή δεν αφορά την ε, ενοποιημένη βάση. Είμαι ερκοντός λογιστής και είναι σταυρός αυτός τον οποίο φέρω και έχω να σας πω το εξής, ότι πρόκειται για το CCATB, δηλαδή πρόκειται περί και όχι ενοποιημένων στοιχείων. Αυτό είναι η πρόταση και οι λογαριασμοί κάθε χώρας ε, προσαρμόζονται για την φορολόγηση. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό οδηγεί σε μια ενοποίηση και ανάλογη φορολόγηση. Οπότε τώρα φεύγουμε τη φορολογία και πάμε στη λογιστική και ο καθένας διαλέγει διαφορετικά λογιστικά πρότυπα για την κάθε θηγατρική της εταιρεία ανάλογα για το τι θα γίνουν με τα κέρδη, που θα αποκριβούν, που δεν αναγνωρίζονται ως τι αυτά κλπ. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός, οπότε αν δεν έχουμε κάποιο είδους συνεπή, συνεκτικά, λογιστικά πρότυπα που να έχουν επίσης σχέση με ε, την ε, αναφορά με την κοινοποίηση χώρα δεν μπορεί να έχουν και εσείς Θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ενιαία πρότυπα. Έτσι να λειτουργεί η λογιστική και να έχουμε ένα αποτέλεσμα από όλα αυτά το οποίο είναι χρήσιμο σαν μπούσουλας. Και ε, το IFRS λέει ότι αυτό δεν βοηθάει. Λέει ότι θα πρέπει οι λογαριασμοί να χρησιμοποιούνται για την φορολόγηση εάν υπήρχε ενίο σετ λογαριασμού, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τα ενία και να προχωρήσει προς τέτοια κοινά πρότυπα κοινοποίησεων των στοιχείων. Άρα να υπάρχουν ε, πρότυπα για κάθε χώρα και το IFRS. Και αυτό θα ήταν πολύ καλό για τις επιχειρήσεις. Μία βάση μία αντίληψη, μία νοοτροπία και όλα αυτά να είναι κατανοητά γιατί οι περισσότεροι λογιστές καταλαβαίνουν ελάχιστα από το τι ισχύει σήμερα. Και γι' αυτό υπάρχουν όλα τα προβλήματα για αυτές τις πιστοτικές κάρτες που προσφέρουν μηδενικό τόκο. Επομένως, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, από τα πιο στοιχειώδη να υπάρχουν οι σωστοί λογαριασμοί που δεν ισχύει σήμερα. Οπότε μόνο από αυτές τις βάσεις μπορούμε να προχωρήσουμε προς ε, κοινή ειδοποιημένη βάση και όχι προς ε, σωρευμένες ε, βάσεις. Και έτσι θα έχουμε φτάσει σε κάτι το κατανοητό για τις ΜΜΕ και για όλους. Άρα έτσι θα έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σύστημα που θα καλύπτει και την αναχώρα κοινοποίηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Brian Hayes για το ΕΛΚ, πρώτος ομιλητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές για το δεύτερο αυτό κομμάτι Συζήτηση Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσει του στο τελευταίο που είπε ο κύριος Μερφή. Έκλεισε για ένα συνεπές σύστημα λογιστικό στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν έχουμε μια ιστορική αγορά και πρέπει ε, να έχει κανείς μια επαγγελματική δραστηριότητα σε μια νέα αγορά, Προφανώ και πρέπει να υπάγεται στι ίδιε προδιαγραφέ με του άλλου. Αλλά σας σα ρωτήσω το εξή. Υποθέσουμε ότι ο κύριο Δεράντ Τραμπ, νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, που μα είπε ότι έχει την πρόθεση να μειώσει την φορολογία των επιχειρήσεων για τις ΗΠΑ. Όντως το πράξη. Τι συνέπειες θα έχει αυτό για τους Ευρωπαίους. Γιατί ένα επιχείρημα το στην είναι ότι καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική την Ευρώπη και ότι θα φύγουν επιχειρήσεις. Θα ήθελα τις παρατηρήσεις σας και δη δημοσία. Ε, δεύτερη ερώτηση. Στη συζήτηση για τους χαμένους και τους κερδισμένους. Εάν ένα κρατός μέλος σκεφτόταν ακόμα και, να, και το ενδεχόμενο να περάσει το σύστημα αυτό, τι συνέπειες έχει αυτό ως προς τα φορολογικά του έσοδα. Και εσείς το είπατε ότι ένα ποσοστό φορολογικής εισφοράς για όλη την Ευρώπη αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Εμείς στην Ιρλανδία έχουμε 15% έσοδα φορολογικά από τους ε, φόρους των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Και άρα σε μια περίσταση κατά την οποία δεν θα υπήρχε η, οικονομική, ε, η αξιολόγηση οικονομικών συνεπειών εν χώρα. Μήπως τελικά αυτό μήνε, ε, σήμαινε αποτυχία των φορολογικών συστημάτων και καταρρευσή τους. Για τους δύο δε ομιλητές. Μια και ο κύριος Μοσκοβησίπε είπε να προχωρήσουμε σε μια βάση και μετά στην ενοποίηση κτλ. Σταδιακά. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Εσείς τι πιστεύετε. Ευχαριστώ ο Πολ Τάνγκ, συζητητής μας από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις και ομιλίες σας. Με ενδιαφέρει το πώς βλέπετε την ιδέα της αγωγής της κοινή ενοποιημένης βάσης ε, φορολόγηση επιχειρήσεων. Θεωρείτε ότι θα περιορίζει την φοροαποφυγή εν γέννη. Η δική μου άποψη είναι ότι ουσιαστικά γίνεται μεταφορά κερδών επί χάρτου. Το τρίτο C, το consolidation, η ενοποίηση, αφορά συγκεκριμένους και αυτού παράγοντες, κεφάλαιο, πωλήσει κτλ. Μήπως μπορέσουν ε, λοιπόν εκμεταλλευόμενοι αυτό το νέο σύστημα οι φοροδιαφεύγοντες ε, για να εκμεταλλευτούν ένα τεχνητό φορολογικό ανταγωνισμό. Και μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και ένα ελάχιστο ποσοστό φορολόγηση. για να μην επικρατήσει ο τεχνητός φορολογικός ανταγωνισμός. Δεύτερον, άειλα αγαθά, άειλο ενεργητικό. Τώρα έχουμε βέβαια τις τιμές μεταβίβασης ως πρόβλημα οι οποίες θα πρέπει να είναι υποτεθεί αγορές τιμές, αλλά τι σημαίνει αγοραία τιμή, ιδιαίτερα σε ενδομιλικές συναλλαγές. Ιδιαίτερα λοιπόν το θέμα τίθεται για το άειλο ενεργητικό. Η Επιτροπή επέλεξε να μην περιλάβει το άειλο ενεργητικό. Εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο νέο σύστημα, όπως κάποιοι προτείνουν τους συναδελφούς. Ή πιστεύετε ότι πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσετε το ζήτημα των τιμών μεταβίβασης. Και ότι είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί και να αξιολογηθεί ποσοτικά, σε τιμέ δηλαδή, το άειλο ενεργητικό. Άρα θα πρέπει να το αφήσουμε αργότερα. Ευχαριστώ. Και ECR τώρα, καθηγητή Λούκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρέπει να πω ξεκινώντα ότι με απογοητεύει η ανταλλαγή απόψεων εδώ, διότι ακούω πολλά έτσι, παρατηρήσει, παρατηρήσεις, πολιτικές θέσεις λιγότερο. Και νομίζω ότι με τέτοια ακρόαση θα έπρεπε περισσότερο να στραφεί στην ουσία μείον εκτήματα πλέον εκτίματα του συστήματος που προτείνεται για την κοινωνιοποιημένη βάση φορολογίας φορολογίες επιχειρήσεων. Ε, τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε τρίτα κράτη. Να μου πείτε το εξής λοιπόν. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, να αντιδράσουν οι επιχειρήσεις αποσυρώμενες, αποχωρώντας προς τρίτες χώρες, ώστε να αποφύγουν τη φορολογία με βάση την αρχή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας επιχειρήσεων. Ή μπορούμε να εισαγάγουμε στο σύστημα κάποια προσκόμματα που δεν θα τους το επιτρέψουν αυτό, ώστε όποια αξία παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αποφεύγει τη φορολόγηση με βάση την κοινωνιοποιημένη φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Και επίσης βλέπω ότι υπάρχει μια διτή προσέγγιση, η δυνατότητα προσέγγισης, είτε μέσω των τρίτων κρατών να γίνονται οι μεταβιβάσεις, οι, οι, ε, μέσα αυτές μεταβίβασης, γίνονται ομιλικές ε, συναλλαγές, είτε η στάθμη συνυπολογίζεται και η στάθμιση θα στα τρίτα κράτη, είτε διαφορετικά να υπολογίζεται ένα τεκμήριο λίγο πολύ κατανομής κερδών με βάση μια αρχή στην οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε. Πάλι όμως με αντιμετώπιση του προβλήματος της διπλής φορολόγησης εισοδήματος που θα έπρεπε να επιληθεί. Πώς θα γίνει λοιπόν η κατανομή των φορολογικών ή φορολογητέων καλύτερα εισοδημάτων. Όταν μάλιστα έχουμε κράτη με τα οποία δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, φερρυπίν, φορολογικές, φορολογικούς παραδείσους της Καραϊβικής. Ε, πώς θα γίνει λοιπόν αυτό να αποφεύγεται η διπλή φορολογία. Thank you very Peter Κοιτάξτε, έχω κάποιες ερωτήσεις προς την κυρία Λατκο Κομουλάινεν. Το όριο των 750 εκατομμυρίων ευρώ το θεωρείτε πολύ ψηλό. Θα θέλατε να περιοριστεί, να πάει στα 40 εκατομμύριο ευρώ πολύ. Είδατε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Ποιες εταιρείες θα το από αυτό το όριο, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν κινούνται απαραίτητα σε πολλά κράτη-μέλη πάνω από ένα κράτος μέλος και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα προσπαθήσουν να φοροδιαφύγουν. Μήπως έχει αρνητικές συνέπειες, το έχετε υπολογίσει αυτό. Στο προηγούμενο πάνελ συζητήσαμε δύο θέματα ε, βασικά. Αυτοί που κερδίζουν και αυτοί που χάνουν από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το CCCTB και ενδεχόμενη μετεγκατάσταση που θα είναι αποτέλεσμα της χρήσεως του συστήματος. Το έχετε συζητήσει αυτό στις συνεδριάσεις σας. Έχετε κάποιες απόψεις επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Μετ Κάθε για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ερώτηση. Κάτι που σχολιάσατε και οι δύο. Ο ρόλος υποβολής εκθέσεων για τα δημοσιονομικά στα πλαίσια του CCCTB θεωρείται ότι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες για τα φορολογικά λογιστικά, πάνω στο οποίο θα βασιζόταν ένα ομοιόμορφο σύστημα φορολόγησης. Η ETUC και το έγγραφο τοποθετήσεως για το CCCTB ζητεί σύγκληση λογιστικών κανόνων. Ο Ρίτσαρτ ανέφερε προηγουμένω ότι τα πρότυπα υποβολή εκθέσεων όπως το IF ε, δεν μπορούν να προσεγγίσουν στα το θέμα. Λοιπόν, μπορείς Ρίτσαρντ να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Τα συμπεράσματα που ανέφερες τις εκθέσεως Πρέμ Σέκαν είναι σωστό το όνομα ή να αναλύσεις το άλλο που ανέφερες. Στάθμιση της εργασίας, πωλήσει αναπροορισμό και μήπως αυτού του είδους ο υπολογισμός μπορεί να αποτελέσει δικείμενο κατάχρησης. Τι εννοείς, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. I hope now I have the right list for... Ε, πράσινη. Σφιν Γκίγκολτ. Σβεν Γκίγκολτ. Το πιάσατε, πρόεδρε, ωραία. Ευχαριστούμε καταρχάς, ευχαριστούμε Ρίτσαρτ για το σχετισμό που έκανες με τους λογιστικούς κανόνες και με το διάσπαρτο τοπίο. Αν επιτρέπει ο Πρόεδρος, θα ξέρω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού, διότι θέσατε κάτι πολύ θεμελιώδες. Ε, συζητούμε τα εθνικά πρότυπα, τα λογιστικά και το IFRS. Εμάς δεν μας ικανοποιούν ε, τα πρότυπα του ISB μέτρα το Λονδίνο. Η πρότασή σας είναι πολύ ευρωπαϊκή προερχόμενη από Βρετανία και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ξέρω επίσης και κάτι άλλο. Ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά τις βασικές παραμέτρους που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως όσον αφορά τα όρια που έχει θέσει για τα μεγέθη και τις πολύ γενναιόδορες διατάξεις όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των στοιχείων ενεργητικού έναντι του χρέους, του συνολικού ενεργητικού έναντι του χρέους. Ακούσατε τον φιλικό Ιρλανδό συνάδελφο και θα καταλάβατε κάτι. Δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη ξεκινούν τακτικισμούς για να κολλησιεργήσουν. Σε εθνικό επίπεδο τα λέμε πιο ξεκάθαρα από το ευρωπαϊκό. Ποιο θα ήταν το όριό σας. Πόσα κράτη-μέλη χρειάζονται για να γίνει λογικό αυτό το σχήμα. Δεν είναι 28-27 κράτη, 29 όπως προτείνατε ή λιγότερα. Ποιο είναι το κατόφλιο το οποίο θα ήταν λογικό για την όλη προσπάθεια για το εγχείρημα. Ευχαριστώ Σβέν. Δεν βλέπω κάποιον άλλον που να ζητά το λόγο στη δικασία Catch the Eye. Πάμε στα μέρη του πάνελ. Πριν πάμε όμως εκεί, θα αναθέσω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρο Νίτελ Μάια. Στην κάτια λέγεται είναι όμως θα δώσω το λόγο πριν φύγω. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις τόσο αξιόλογες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν φοιτητρία νομική στην Φιλανδία και έμαθα την αρχή ε, που διέπει, τι αρχές που δουλεύει την φορολογία ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα, να υπάρχει σαφήνεια, θα πρέπει να υπάρχει απλώτηση στους κανόνες που διέπουν το φορολογικό δίκαιο. Αυτές είναι οι βασικές αρχές που ακόμα ισχύουν. Πρώτα, πρώτα. Πρώτη ερώτηση. Η ETUC. Και είναι πολύ σημαντική σε αυτές τις φάσεις, αλλά το είπαμε αυτό ήδη. Το είπαμε. Η TUC ζητεί ταχεία υλοποίηση, ολοκλήρωση αυτής της δεύτερης φάσης της STB. Δεν είναι σαφές προς το παρόν το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή, για την δεύτερη παρατήρηση. Θέλουμε να υπάρχει ελάχιστο συντελεστή για τι εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούν τα μέλη μας προ τούτο. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Και έτσι θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις να ψάχνουν πού είναι πιο χαμηλή φορολογία γύρω-γύρω. Ο τρίτος κύριος που έλαβε κατά σειρά το λόγο ανέφερε για τις τρίτες χώρες. Είπε ότι τον απογοητεύουν τα όσα είπαν, αλλά για τα μέλη μας, το ETUC που τα μέλη μας έρχονται από τις δικές σας χώρες, δεν τους νοιάζει εάν ξεκινά όλα αυτά από το CCTV ή αν προέρχεται από κάποια άλλη νομοθετική πρόταση το αποτέλεσμα ο κόσμος νοιάζεται για το αν θα πληρώνει ή δεν θα πληρώνει φόρους. Θέλουν δικαιοσύνη σε αυτό. Να είναι σαφής οι κανόνες. Όπως ο κόσμος πληρώνει φόρους, θέλουν και οι εταιρείε να τους καταβάλουν. Κάτω έχουμε και τις λεπτομέρειες, αλλά εδώ δίπλα μου ο καθηγητής θα σας εξηγήσει τα τεχνικά σημεία. Είναι σημαντικό, επομένως, έτσι να δούμε το πράγμα. Έτσι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει θεμέλια δίκαιους κανόνες. αυτά που μου λέγανε στην νομική οι καθηγητές. Τώρα, ο τέταρτος ομιλής από τους φιλελευθέρους. Δεν μιλάμε για όλες τις Ε, ναι, είναι καλή ερώτηση. Ναι, αυτό είναι σημαντικό και δεν έχει παλιότερα αντιμετωπιστεί. Όλα αυτά τα θέματα για έρευνα και ανάπτυξη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει και τα σχετικά κίνητρα. Και εμείς αυτό θέλουμε, ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εταιρείε να υπάρξουν νέε ιδέες, να υπάρξει έρευνα και ανάπτυξη. Ε, με αυτό είναι. Και του CCTV, καλύπτει και τα σχετικά κίνητρα. Από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, ο πέμπτος ομιλητής που μίλησε για την προτυποποίηση, τα ξέρει καλύτερα αυτά ο καθηγητής Μέρφυ. Έχει περισσότερη εμπειρία τόσο ώστε να σας πει τα σχετικά. Αλλά όπως σωστά είπατε, εμείς είμεθα υπέρ, υπέρ των επιχειρημάτων που ήδη πρόταξε ο κύριος Μέρφυ, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, Είναι λογιστικά πρότυπα. Αλλά και ο κύριος από τους Πρασίνους έθιξε το θέμα, τον, ε, το, το λογιστικό. Και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος και την τρώτο λόγο ή στον καθηγητή Μέρφυ για πέντε λεπτά. 13 ερωτήσεις έχω σημείωσα, οπότε θα πρέπει γρήγορα να σας τα πω σε πέντε λεπτά. Έχουμε πρόβλημα με την φορολογικό ανταγωνισμό, υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι και έχουμε και άλλη μια ερώτηση πιο κάτω, κατά πόσο αυτό οδηγεί σε τεχνητή μετακίνηση με την κατάσταση εταιρεών και εθνικών. Μα ποια είναι η ουσία, ποια είναι η οικονομική ουσία τη φορολογική, τι συμβαίνει τώρα. Είναι ότι οι εταιρείε αποφασίζουν ε, επί τη βάση του που έχει πιο εκπαιδευμένου, που έχει καλέ υποδομέ, που υπάρχει καλύτερο δίκαιο, που θα έχουν υψηλότερη ποιότητα από διάφορε απόψει και έτσι αποφασίζουν πού θα αναπτύξουν τη δραστηριότητα, που θα βάλουν του υπαλλήλου στο πρόβλημα. Με το ενωτερικό φόρο είναι ότι τα κέρδη δεν είναι εκεί που αναπτύσσεται η δραστηριότητα. Και αυτό είναι το, η κοινή ενωπημένη βάση. και ο τρόπο εφαρμογή είναι ότι θα ληφθεί υπόψη ακριβώ πού γεννάται το κέρδο. Και ο Μπάφετ έλεγε ότι κανεί δεν θα πει όχι σε ε, σε μια χώρα θα αρνηθεί να, να κερδίζει επειδή εκεί πέρα υπάρχει εφορολογία. Επομένω, δεν θα μετακινείται τεχνητά ο κόσμο. Τώρα, κατά πόσο έχουμε κερδισμένου, χαμένου, ναι, αν έχουμε χαμένου θα είναι οι χώρε οι οποίε σήμερα δεν εισπράττουν του φόρου όταν μπορούν. Μιλάμε για 13 δις περίπου ή για άλλο λόγο τελικά δεν ε, εισπράττουν του φόρου. Ε, α αλλάξουν. Τώρα χρειάζεται η ενωπημένη βάση ή θα πρέπει να μην είναι ενωπημένη. Θα πρέπει να είναι. Προ τα εκεί θα πρέπει να πάμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε κάτι μεσοδέζικο. Θα είναι πιο δύσκολη φορά αποφυγή αν υπάρχει αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Και τι, τι, τι είναι η υποβολή των στοιχείων ή το CCTV ένα μεγαλύτερο, πιο πολλά αποτελέσματα θα φέρει υποβολή στοιχείων ανά χώρα. Εγώ κάτσε και έχω συνομιλήσει με προσώπους ε, εταιριών, συγκεκριμένα στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και μου είπαν ότι μπορούν πολλά να καταφέρουν ε, με την υποβολή στοιχείων ανά χώρα. Και τώρα θεωρούν ότι σύντομα πρόκειται να προχωρήσει η Ευρώπη σε αυτό το μέτρο αλλά τελικά θα αλλάξουν και οι εταιρείε και οι αρχές την συμπεριφορά και θα υπάρξει συμμόρφωση. Τι γίνεται με τα άειλα. Τα, τα άειλα δεν έχουν αξία. Μόνο εάν τα δημιουργούν πραγματικοί άνθρωποι μπορούν να τα συντηρήσουν, να τα διατηρήσουν. Δεν υπάρχει καμία αξία στα άειλα παρά μόνο εάν επιδέχονται μεταβίβαση, πώληση. Επομένως ε, το θέμα είναι η πώληση. Οπότε γι' αυτό και θα καλύπτονται όλα τα άλλα άγαθα, όλα τα άλλα στοιχεία ενεργητικού που τώρα ε, υπολογίζονται στον φορολογικό προγραμματισμό. Και υπάρχουν και φυσικά μηχανισμοί για τη χειραγώγηση των κερδών. Τώρα κάποιο καθορισμένο κράτος μέλος θα αναλάβει την πατρότητα του μέτρου αυτού. Μπορεί να οριστεί. Ιδάλλως, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αναθέσει στις φορολογικές αρχές. Και έτσι θα έχει τη σχετική ευθύνη αυτή η αρχή. Ιδάλλως όποιος και όποια εταιρεία δεν υποβάλλει τα σχετικά στοιχεία δεν θα μπορεί να ασκεί εμπορία τι γίνεται με τις πλασματικές τιμολογήσεις, με μόνο μεταβίβαση κλπ. Ε, αυτό θα, θα απαιτούσε και χρειάζεται υποβολή στοιχείων σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ΣΑ, όπου και εκεί έχω υπηρετήσει και έχω ακόμη επαφή, εξετάζει το κατά πόσον μπορεί να ρυθμίσει αυτό το θέμα των τιμών μεταβίβασης επί τη βάση του πώς χωρίζονται και κατανέμονται τα κέρδη από τις εταιρείες. Άρα προς τα εκεί πάμε. Συμφωνώ με τα χαμηλά κατόφλια. Δεν ξέρω καν αν αρκούν 40 εκατομμύρια. Χρειάζονται τα στοιχεία. Δεν ξέρω αν για τις πολυεθνικές αυτό κολλάει. Πωλήσει αναπροορισμό μπορούν κάποιοι συνεργάτες να το κάνουν αυτό Μπορεί αυτό να το κάνει και κάποιος στα νησιά Κέιμαν. Μπορεί να υπάρχει franchising ή να μην υπάρχουν πωλήσει προς τρίτους. Αυτό βέβαια είναι στρέβλωση. Είδατε τι είπε ο Τραμπ. Αυτό είναι κίνδυνος και θα κηρυχθεί παράνομο. Όπως χρειάζεται και η απασχόληση ανά πρόσωπο και ανά αξία. περισσότερες μεγάλες εταιρείες, προς μικρές εταιρείες, δεν κάνουν έρευνα και ανάπτυξη που εκπίπτει. Δεν έχουν το κεφάλαιο. Άρα να μην προσποιούμεθα ότι αυτό το μέτρο θα ωφελήσει τις ΜΜΕ. Ας τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά, τα οποία βέβαια συνεχίζουν να ωφελούν τις μεγάλες εταιρείε, αλλά μία πολυεθνική θα πρέπει να συμμορφωθεί με την ενωπημένη βάση Αλλιώς θα παραβιάζει τους βασικούς λογιστικούς κανόνες. Οπότε το πρόβλημα είναι πάλι τα λογιστικά. Γιατί κάποιος δεν έχει λογιστικά βιβλία, ε, τότε αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τις φορολογικές αρχές. Νίτερ Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα παρακαλώ την Επιτροπή. Ποιος θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση. Έχετε λίγα λεπτά χρόνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήταν χρήσιμο όντω να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που μας αφορούν. Είναι και χαρά μου βεβαίω. Μα ε, ενθαρρύνει πολύ αυτή η συζήτηση, μας ε, προσφέρει τεράστιο υλικό για τη σταθεροποίηση της ε, πρότασης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και βεβαίως πολύ ευχαριστώ να συνεχίσω τις συνομιλίες με κάποιους από εσά. Ε, για τέσσερα σημεία καταρχάς. Ευελιξία, στοιχείο ευελιξίας. Αυτό που κάνουμε είναι να προτείνουμε μία πρόταση για εναρμονισμένη φορολογική βάση επιχειρήσεων. Όντως, και πολλές είναι οι επιχειρήσεις που το καλωσορίζουν αυτό, προτείνουμε ένα πολύ σταθερό σύστημα σύστημα το οποίο δεν θα εκθέσει τις επιχειρήσεις μας στο σύνολό τους σε μια διαρκή ετήσια αλλαγή του ε, φορολογικού τους περιβάλλοντος. Ε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ευελιξία έχει ε, ρόλο στο εξής, ότι είναι υποχρεωτική σε σχέση με ένα συγκεκριμένο όριο το βάζουμε το όριο αυτό στο τραπέζι. Καταλαβαίνω τα ερωτηματικά που λένε γιατί αυτό το όριο έχει κάποιο άλλο, αλλά πάλι είναι η Επιτροπή ανοιχτή για συζήτηση. Πάντως το ερώτημα είναι να έχουμε την ευελιξία για μικρότερες επιχειρήσεις, ώστε αυτές να μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να, να υπαχθούν ή όχι, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Περισσότερη ευελιξία δηλαδή για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Και επίσης το στοιχείο της, ε, των λογιστικών λογαριασμών. Βεβαίως είναι δύσκολο να έχουμε συστήματα για την ε, φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων, όμως ε, μην κατηγορείτε το CCTB ότι δεν κάνει αρκετά για την φορολογική καταγραφή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε το CCTB είναι, με το νομοθέτημα, είναι να μην αφήνουμε στα χέρια των μη κρατικών φορέων την απόφαση για το πώς θα γίνει η φορολογία. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η πρόταση, ποια ε, είναι τα φορολογητέα κέρδη για να μην μείνει αυτό σε ιδιωτικά χέρια αλλά στα χέρια των δημόσιων, ε, των κρατικών αρχών του νομοθέτη βασικά. Επίσης νομοθεσία και άρθρα πολλά μας δείχνουν ε, ποια είναι η πολιτική πραγματικότητα στην Ευρώπη και δεν είναι, που δεν είναι η πρόθεσή μας να περάσουμε σε ένα ελάχιστο συντελεστή φορολογίας. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Μπορεί κανεί λοιπόν να προτείνει ένα τέτοιο επιχείρημα, αλλά η πολιτική πραγματικότητα και η αποτελεσματικότητα τη συζήτηση του που θέλουμε να προχωρήσουμε, προ τα που θέλουμε να πάμε, είναι ακριβώ αυτό της διαφάνειας, κατά ε, της φοροαποφυγής και του θετικού φορολογικού σχεδιασμού και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη με βάση τη διαφάνεια μπορούν να επιλέξουν δεν αληθεύει σε αυτό που ακούστηκε τώρα από τον Ρίτσαρτ, το άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν ε, αντιμετωπίζουμε το ε, ενεργητικό. Όχι. Μπορεί να μην αναφέρεται ρητά, αλλά όταν είναι μέσα σε έναν όμιλο, τότε και εκεί θέλω να ακούσω τι έχει να πει ο Ρίτσαρτ, χρειάζεται κάποιος τρόπος να υπολογιστεί. Δεν, ε, δεν πέφτει από τον ουρανό το άϊλο. Επομένως πρέπει να δούμε με τι κόστος, με τι κέρδος κτλ. Παράγεται το άϊλο αυτό. Ενεργητικό. Πάντως υπάρχουν συστήματα τα οποία λειτουργούν πολύ καλά, πολύ αποτελεσματικά. Και γι' αυτό νομίζω ότι και για να ολοκληρώνω το τελευταίο και πολύ σημαντικό σημείο, η ιστορία, η σχετική η συζήτηση σχετική με τους χαμένους και τους κερδισμένους. Θα συμφωνήσετε πιστεύω ότι δεν είναι το σύστημά μας ε, πρόσφορο για να υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Δεν προξενεί κερδισμένους και χαμένους. Αντιθέτως, ε, επιτρέπει τη σύγκληση προς μια κατεύθυνση προς ένα σύστημα το οποίο να επιτρέπει στον καθένα την προσαρμογή. Και αυτό είναι το πνεύμα μας. Με αυτό θα μπούμε στη φάση των διαπραγματεύσεων για το CCTB. Στοιχεία υπάρχουν, είμαστε απόλυτος διαφανείς για το τι σημαίνουν τα στοιχεία αυτά. Γιατί είναι στοιχεία που προέρχονται από ε, μοντέλα και θα συμφωνήσω ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Πολλές φορές βλέπω διάφορες μελέτες ε, να ανακοινώνονται στον τύπο, αλλά δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, λέει, γιατί δεν μπορούμε να, να τις καταστήσουμε δημόσια γνωστές και εμείς δεν είμαστε θέση να αντιπαραβάλλουμε τα στοιχεία που έχουμε από το ένα κράτος στο άλλο. Ε, εκεί θα ήθελα να μπορούμε να διευκρινίσουμε ποιοι είναι οι χαμένοι και οι κερδισμένοι και να κάνουμε τη σχετική προσαρμογή ώστε να είναι κοινά αποδεκτό αυτό. ώστε να είναι αποδεκτή αυτή η πρόταση τελικά στο τέλος των πραγματεύσεων. Άρα χρειάζεται μία βάση που θα μας δίνει όλα τα στοιχεία, τα απαραίτητα για την πρόθεση της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούν οι συγγητές σας, ο Πολ Τάνκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, uh, Ευχαριστώ εκ νέου για αυτά που μας είπατε. Πολλά σχόλια ακούστηκαν. Προσπαθώ να δω πώς θα τα προσεγγίσω όλα αυτά. Από τη συζήτηση είναι σαφές ότι όλοι βλέπουν τα τρία αυτά C ε, μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα. Δεν άκουσα κάποιον άλλον να πει ότι θέλει να αλλάξουμε κάτι ή να διαχωρίσουμε τα τρία C. Σαφέστατο το μήνυμα. Όπως είπα και στην αρχή, πιστεύω ότι το CCCTB έχει δυνατότητες να είναι ένα πολύ σύγχρονο φορολογικό σύστημα. Αν δείτε ότι αυτό που κάνει και Τρόμπ είναι κάπως οπισθοδρομικό. Ακολουθεί εδαφική προσέγγιση. Το πρόβλημα με, με το άειλο ενεργητικό ή τις μεταφορές ενεργητικού μεταξύ επιχειρήσεων. Είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί με αυτό το τύπο κατανομής να θεσπίσουμε ε, νέους κανόνες που θα ισχύουν πάντοτε. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Θα πρέπει όλα αυτά να μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και επίσης τι γίνεται και με τα κέρδη ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. όλα αυτά είναι υπέρ των μικρομεσών επιχειρήσεων, δημιουργούνται ισότιμες συνθήκες, αυτό είναι σημαντικό. Επιτρέπουμε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρόκειται να κινηθούν διεθνώς, αυτό θέλουμε, να μεγαλώνουν οι μικρές επιχειρήσεις, να τις υποστηρίξουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και έτσι γίνεται απλούστερο το φορολογικό σύστημα. Είναι απλό και βανάγνωστο αυτό που προτείνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί και κομπλιμέντο. Άρα, είναι η πρώτη φορά που διεξήχθη συζήτηση, την εκτιμώ, σημείωσα πολλά σχόλια. Διότι τι θέλουμε στο τέλος. HGI, τι γίνεται με το οικονομική κρίση κλπ. Η σταθερότητα είναι κάτι που ε, τίθεται σαν θέμα. Τι θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος. Έχουμε μια πρόταση που να την στηρίζουν. Να τη στηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οργανώσεις των εργοδοτών. Και ακόμα και οι χώρες ε, που είναι πολύ διστακτικέ, που είναι οι μικρότερες να το στηρίξουν. Πρέπει αυτή η πρόταση να γίνει τέτοια, ούτως ώστε να είναι μια προσφορά που κανείς να μην μπορεί να την αρνηθεί. Αυτά και ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή του συζήτηση. Ευχαριστώ Πολ. Ο Αλάν Λαμασούρ, Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ με τη σειρά μου, λέει ο Λαμασούρ, όλους τους ομιλητέ. Δεν έχω την ίδια άποψη όπως ο Μπεντ Λούκε, ο συνάδελφος. Μιλάμε κάπως γενικά, αλλά η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η συνεισφορά των μελών που μίλησαν ήταν ε, πολύ καλές. Σημείωσα δεόντως την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση περί των αήλων ε, στοιχείων ενεργητικού. Όσον αφορά την ανάλυση ότι οι υπερβολικές μειώσεις που προτείνονται στα πλαίσια του φόρτου κεφαλαίων για να μην υπάρχει μεροληψία όσον αφορά κάποιες επιχειρήσεις και κάποιες χώρες ήταν ενδιαφέροντα για την ευελιξία Το βλέπουμε σε όλα τα κείμενα που αφορούν τις δραστηριότητες οικονομικές και τις τραπεζικές που συζητούμε εδώ. Αλλά υπάρχει δυσκολία όσον αφορά αυτό. Η διάρκεια των διαδικασιών για την, τροπολογία, για την τροποποίηση μιας οδηγίας όταν έχει εγκριθεί αυτή. Και πιο γρήγορα μπορεί να κινηθεί κανείς σε εθνικό επίπεδο και είναι κάτι πιο ευέλικτο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο της ευελιξίας. Δύο σχόλια. Έχω δύο ερωτήσεις. Το κατόφλι πρώτα απ' όλα. Η δεξιά λέει μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, χρησιμοποιούμε αυτό το όριο ε, των 150 εκατομμυρίων ευρώ στις αναχώρα εκθέσεις. Σύμφωνα με προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΟΣΑ η αριστερά λέει όσο πιο χαμηλό το κατόφλι τόσο το καλύτερο. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κατόφλι όμως. Το χρειαζόμαστε. Διότι πρέπει να διαλέξουμε. Έχω μια πολύ υπεραπλουστευμένη προσέγγιση και ένα σχόλιο. Εάν το σύστημα που θέλουμε να θεσπίσουμε αποτελεί πρόοδο. Εν τη αυτή περι, ε, περιπτώσει γιατί να περιορίσουμε την πρόοδο στις πολυεθνικές. Θα έχουν δυνατότητα εθελοντική συμμετοχής οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό περιπλέκει πολύ υπερβολικά τα πράγματα. Ή το σύστημα που θεσπίζουμε από την άλλη θα είναι επιβαρυντικό για τι επιχειρήσει. Σε αυτή περιπτώση, γιατί να το δημιουργήσουμε. Θέλουμε πρόοδο, αυτό είναι προφανέ. Πρόοδο που συνεπιφέρει τις λιγότερες επιπλοκές εν πάση περιπτώσει υπάρξουν επιπλοκές διότι θα μεταμορφώσουμε σε κάθε χώρα ένα φορολογικό σύστημα για τη φορολόγηση εταιριών και θα γίνει κάτι άλλο είτε άλλο εθνικό σύστημα ή ένα άλλο κοινό σύστημα που θα καλύπτει πολλές χώρες, ιδεοδός και τις 27. Θα πρέπει με σοβαρότητα να μελετήσουμε τη δυνατότητα να εφαρμοστεί το σύστημα στο σύνολο των επιχειρήσεων και όχι μόνο σε εκείνες που έχουν μια δραστηριότητα σε πολυεθνικό επίπεδο. Εξάλλου έτσι λειτουργεί και στο Ομοσπονδιακό Σύστημα των ΗΠΑ για κάποια χρόνια θα υπάρξει περίοδος κάπως περίπλοκη για όλους, αλλά μία φορά θα συμβεί αυτό. Θα κρατήσει δύο, τρία, τέσσερα χρόνια ε, το πρόβλημα. Και αφού θα γίνει η προσαρμογή, όλα θα είναι εντάξει. Διαφορετικά. Αν έχουμε ένα σύστημα που μόνο οι εταιρείε πάνω από κάποιο κατόφλι, όποιο και να είναι αυτό, θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά το σύστημα και οι άλλε επιχειρήσει μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά, αυτό θα ανοίξει νέα κενά και θα, ε, γίνουν, θα υπάρξουν άλλα προβλήματα προσπάθειες βελτιστοποίησεως. Δεν έχω απάντηση, πρέπει να τεθεί το ερώτημα. Τελευταίο σχόλιο τώρα. Το θέμα των winners και losers, ε, losers είναι ψευδές πρόβλημα. Ποιος, ποιοι θα είναι οι winners, ποιοι θα είναι οι losers. Αν μπορεί μια χώρα να πει ότι χάρη στο CCCTB Τελικά οι επιχειρήσει που είναι κατεστημένε σε εμά θα πληρώνουν λιγότερου φόρου από πριν. Αυτή η χώρα τι θα είναι, winner ή loser από πλευρά δημοσιονομική. Μπορεί να χάσω κάποια χρόνια, αλλά θα προσελκύσουν ξένε επενδύσει. Μην χρονοτριβούμε κολλώντας εδώ. Πιστεύω ότι δεν είναι πραγματικό πρόβλημα, είναι ψεύτο πρόβλημα αυτό. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ όλους που μιλήσαμε και συζητήσαμε αυτό το δίωρο. Έξοχη ε, έναρξη συζητήσεως ενός πολύ σημαντικού θέματος. Θα διακόψουμε και σε τρία λεπτά θα συζητήσουμε το επόμενο θέμα. Dear colleagues, please may I ask you to take seat. We move to uh, point 13. Ο πρόεδρος λέει πάμε στο σημείο 13 της ημερησίας διατάξεως το οποίο αφορά την αξιολόγηση επί των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Mm. Με μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή έχουμε κοντά μας και στην Επιτροπή μας τον κύριο Ζακ Ντελαροζιέρ. Περιτεύουν τα λόγια παρουσίασής του γιατί τη σταδιοδρομία του. Είναι δεμένη με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, ΟΝΕ της Ομοσπονδιακής Ένωσης. Οπότε είναι μεγάλη μας τιμή, είναι ένα προνόμιο να τον έχουμε εδώ. Είναι στέλεχος στην Τράπεζα της Γαλλίας, στο Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο, στην Τράπεζα ε, Περιφερικής Ανάπτυξης και έχει και άλλα αξιώματα πολύ σημαντικά. Και όπως γνωρίζετε είχε το Κέντρο Προβληματισμού για το Τενές Νομισματικό Σύστημα για την Νομισματική Ένωση και μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Ανέλαβε την πατρότητα της φημισμένης έκθεσης για το σύστημα ΕΖΑΣ, δηλαδή τις Ευρωπαϊκές Ευρωπαϊκές Αρχές. Αυτέ οι αρχέ τώρα υφίστανται αυτή την αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία δημοσία διαβούλευση η οποία επεβάλλεται. Είναι κάτι το οποίο το διοικητική πολύ καιρό το κοινοβούλιο γιατί προβλέπεται νομοθετικά μια τέτοια αξιολόγηση. Ιδίω τώρα στους καιρούς του Brexit. πλευρό γεγονός, αλλά επίσης πρόκειται να αποτελέσει και κίνητρο του να προχωρήσουμε εις το μέτωπο της σύγκλησης της εποπτικής λειτουργίας. Οπότε και έγινε αυτή η, διαβούλευση για την αξιολόγηση. Να δούμε την αρχιτεκτονική του συστήματος εποπτείας. Όλα αυτά τώρα συζητούνται. Διάφορες παραλλαγές της δομής αυτής. Και να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχει αποτελεσματικότητα, τι γίνεται με τα θέματα της χρηματοδότησης, οπότε βεβαίως και πρόκειται να εμπλακεί σε αυτή τη διαδρομή. Το Κοινοβούλιο είναι και συνομοθέτης αλλά να δούμε και τι ε, timing προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε τελικά να προχωρήσει αυτή η νομοθετική πρόταση. Μεγάλη μου χαρά Ζάκη, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Επανειλημμένα έχουμε ανταλλάξει απόψεις στο παρελθόν και ανέκαθεν. Με μεγάλη μου χαρά έχω συμμετάσχει αυτές τις ανταλλαγές απόψεων. Είναι τιμή μου σήμερα να σας πω τις σκέψεις μου όσον αφορά την λειτουργία αυτών των τριών εποπτικών αρχών που συγκροτήθηκαν το 2009 τότε που προείδρευα σε αυτή την προσπάθεια. Έχει περάσει μια επταετία έκτοτε. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση, να δούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των φορέων, αυτών των οργάνων για το μέλλον όπου θα πρέπει να δούμε τι ισχύει και σε σχέση με το Brexit. Και στέκει να πει κανεί ότι αυτές οι τρεις αρχές επετέλεσαν έργο αξιόλογο όσον αφορά την αποστολή τους. Πέτυχαν. Πέτυχαν λόγω της ποιότητας του προσωπικού, λόγω της ποιότητας των διοικούντων. Ε, ε, και ήταν κέντρα μεγάλης ικανότητος. Και αυτό και παγκοσμίω. Επίσης ήταν ο ρόλος του κλειδί, ούτω ώστε να έχουμε ενιαία ε, ρύθμιση για αγορές, τράπεζες και ασφάλειες. Ενιαίο κώδικα που, που να διέπει αυτές τις, αυτούς τρεις τομείς. Έχω εδώ μια ολόκληρη ομιλία όσον αφορά τα επιτεύγματα. Αλλά για να είμαι πιο σύντομος και να τηρήσω και το πεντάλεπτο το οποίο μου παραχωρήσατε δεν πρόκειται να αναφερθώ στο πρώτο τμήμα. Εάν θέλετε μπορείτε αυτά να τα βρείτε στο σχετικό κείμενο το οποίο έχει διανεμηθεί. Οπότε θα περιοριστώ στις προκλήσεις και στις νέες εξελίξεις. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εάν θέλουμε να προχωρήσουμε προς πιο αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και πρώτα πρώτα έχουμε το πρόβλημα της αξιολόγησης των μελών των διοικητικών συμφουλίων. Θα πρέπει να υπάρχει μόνο λεπτομερής και εντελεχής ρύθμιση από τι κανονικέ αρχές και όχι αποκλειστικά από τις εποπτικέ αρχές. Κάτι το παράδοξο τώρα έχει ε, τρυπώσει στην λειτουργία αυτών των εποπτικών αρχών. Το λέγαμε και πριν από λίγες εβδομάδες. Να σας πω την άποψή μου. Τι γίνεται τώρα. Μόνο οι εθνικές εποπτικές αρχές συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των εποπτικών αρχών, αλλά όχι οι ρυθμιστικές εθνικές αρχές. Δηλαδή, βασικά τα Υπουργεία Εθνική οικονομίας και οικονομικών. Οπότε είναι κάπως παράδοξο το να ζητεί κανεί από τις ευρωπαϊκές αρχές να εποπτεύουν την θέσπιση νομοθετικών μέτρων. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Η δουλειά των εποπτικών αρχών. Οπότε βέβαια είναι καλή ιδέα να συμμετέχουν οι πολιτικές αρχές στα διοικητικά συμβούλια, αλλά Αλλά εκεί θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ρυθμιστικών αρχών. Γιατί η σημερινή πρακτική έχει πολλά μειονεκτήματα πρώτα-πρώτα. Δεν αισθάνονται πάρα πολύ άνετα οι εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών όταν κάνουν να νομοθετήσουν. Και βέβαια, το πρόβλημά τους είναι όταν ε, τελικά καλούνται να κρυθούν οι υποπτικές αρχές ίδιες και να αξιολογηθούν. Οπότε το να ζητούμε από αυτούς τους επόπτες των ΣΥΠΗΝ να μετέχουν σε αυτά τα διευθυντικά όργανα, ε, τότε αυτό είναι συνταγή ακινησίας. Να, ποια είναι η πρώτη μου παρατήρηση. δεύτερη τώρα, το να δείξουμε μία ματιά στα θέματα της διακυβέρνησης που χαρακτηρίζουν αυτά τα διοικητικά όργανα. Το σημερινό οποίο λέει ότι οι εθνικοί εκπρόσωποι ε, είναι οι βασικοί ρυθμιστέ των όσων γίνεται σε αυτά τα όργανα τα διοικητικά, διευθυντικά. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί μια ευκαιρία οι εθνικές αρμόδιες αρχές μονομερός να προσαρμόζουν κάποιους κανόνες και να προσθέτουν κάποιο είδους τοπικές απαιτήσεις με στόχο να προστατεύσουν τους συμπατριώτες τους είτε είναι καταθέτες είτε είναι εισφαλισμένοι. Οπότε έτσι. Οτιδήποτε γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε αντίφαση με το ζουμί, το σκοπό της υπόθεσης. Και έτσι έχουμε και κατάτμιση σε μεγάλο βαθμό αλλά και έτσι αποδυναμώνεται η χρηματοπιστωτική ενιαία αγορά, όπως και η Τραπεζική Ένωση. Επίσης, έχει υποθεί ότι υπό κάποιες συνθήκες οι πολιτικές αυτές αρχές δεν έχουν μπορέσει να προβούν σε μια συγκροτημένη εφαρμογή των τεχνικών κανόνων και διατάξεων. Αν αυτό το λάβουμε υπόψη, ε, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση. Γιατί έχουμε τις σχετικές ε, κοινωτικές υπηρεσίες, αρχές προτιμώ να τις ε, ονομάζω, όπου το έργο τους είναι να νομοθετούν. Και οι υπότικες αρχές να βλέπουν κατά πόσο υπάρχει ορθή εφαρμογή. Όμως τώρα αυτές οι αρχές είναι χωρίς καμία εξουσία. Είναι τελείως αδύναμες. Δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ε, αποτελεσματική εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. Οπότε, οι υποπτικές αρχές μπορούν να επισημάνουν, μπορούν να ε, διερευνήσουν τις ε, παραβάσεις του δικαίου, το, gold plating, τα, τα παραθυράκια, τις ανεπάρκειες του νόμου, συστημικούς κινδύνους, αλλά δεν μπορούν να ενεργήσουν στη συνέχεια όπως έχουν τα πράγματα σήμερα γιατί δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Αν λίγο το σκεφτείτε θα δείτε ότι να, εμείς έχουμε απονείμεις σε αυτούς τους φορείς την αρμοδιότητα ούτως ώστε να νομοθετούν ε, σύμφωνα με το πρώτο επίπεδο των σχετικών οδηγιών. Από εκεί Ο Όμως αυτοί οι κανόνες αποκτούν, έχουν μόνο θεωρητική αξία. Εάν δεν κάνουν ό,τι πρέπει οι χώρες. Άρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πίεση από τους ομολόγους και ομοτήμους είναι εδώ το θέμα. Όχι, λέγω, δεν ισχύει αυτό. Αυτή η πίεση είναι μια ωραία βρετανική έκφραση. Αλλά δεν ωφελεί για χώρες που αποφάσισαν να αποκλίνουν από την κοινή αντίληψη περί τα πράγματα. Άρα, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα της αρμοδιότητας των κυρώσεων, είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό. Να δούμε τι θα γίνει με την τροπεζική Ένωση, τι θα γίνει με το CMU, τι θα γίνει με τη διαμεσολάβηση τραπεζική, τι θα γίνει με την επίλυση διαφορών μεταξύ των αρχών και πόσο όλα αυτά θα πρέπει να ασκούνται ως επιλογές περισσότερο. Αλλά κυρίως ε, θα πρέπει να δούμε το πόσο θα υπάρξει ανάθεση σε κυρωτικές αρμοδιότητες προς αυτές τις αρχές. Για να μπορέσουμε τώρα να προωθήσουμε το γενικό κοινοτικό συμφέρον, όπως το λέμε, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι τα διαχειριστικά όργανα ε, των πολιτικών αρχών γίνεται να μετασχηματιστούν και να είναι κάτι σαν εκτελεστικά διοικητικά συμβούλια και να έχουν μόνιμα μέλη, τα οποία να μην προέρχονται από τις εθνικές αρχές. Ένα τέτοιο ε, συμβούλιο, όργανο, εκτελεστικές αρμοδιότητες θα είχε σημαντικό ρόλο. Θα είχε αποφασιστικές αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς όπως για δεσμευτική διαμεσολάβηση, για επιτόπου επιθεωρήσεις, ελέγχους και τα μέλη επίσης θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και στα εποπτικά συμβούλια και όργανα και όλες αυτές οι μεταβολές θα έκανε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων πιο αποτελεσματική και πιο συγκεκριμένα πιο ευρωπαϊκή. Τώρα, κάποιες άλλες αλλαγές που θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόδοξες από αυτά που προαναφέραμε έχουν διατυπωθεί από διάφορους ε, των εμπλεκομένων και λένε για το πώς θα πρέπει να είναι κάτι το πιο κεντροκατευθυνόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποιες ε, υποπτικές λειτουργίες οι οποίες αφορούν κάποιου είδους δραστηριότητες ή κάποιου είδους νομικά πρόσωπα που δρούν διασυνοριακά, όπως πούμε να υπάρχει ε, κάποιο είδους καταγραφή κάποιων ε, διαδικασιών ή προϊόντων και άλλοι έχουν πει ότι θα πρέπει να ε, διευρυνθεί το, το τι μπορεί να κάνουν αυτές οι, οι αρχές, η ΟΠΑ και οι άλλοι, και άλλες εποπτικές αρχές, γιατί η ΟΠΑ θα μπορούσε να της ανατεθεί ο σκοπός το να έχει κάποιο είδους κεντρικό εποπτικό ρόλο στην συνεχή εποπτεία κάποιων προτύπων βέβαια αν είχε τους κατάλληλους πόρους προς τούτο και μπορούσαμε να ανατεθούν και άλλες τεχνικές ε, αρμοδιότητες προς αυτές τις αρχές και κυρίως όσον αφορά τους νέους τραπεζικούς κανόνες όσον αφορά το πρωτογενές δίκαιο. Και έχει αποδειχθεί ότι έτσι μπορούν αυτοί να συνεργαστούν με τα τρία θεσμικά όργανα για αυτά τα θέματα. Και όπω και να προχωρήσει περισσότερο και να αναθέσει αυτές τις αρχές και νομοθετικές αρμοδιότητες. Άλλο τώρα, άλλη ιδέα λιγότερο φιλόδοξη αλλά πολύ πρακτική είναι να επιτραπεί σε αυτές τις αρχές να μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να έχουν πρόσβαση εις πληροφορίες αν χρειαστεί. Και μου φαίνεται πάρα πολύ παραδοξικό ότι με την Ένωση των, των, Τραπεζών που υποπτεύει, υποπτεύει την υποπτία των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η EBA ε, έχει κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά την ερμηνεία κάποιων δεδομένων που προέρχονται από κάποιε εκ των τραπεζών αυτών, η EBA δεν μπορεί να κλητεύσει την τράπεζα αυτή και να πει δεν καταλαβαίνω να την εγκαλέσει τη συγκεκριμένη τράπεζα και να πει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορεί, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Την τράπεζα κάποιε χώρε. Πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στι εθνικέ αρχέ. Το βρίσκω λίγο παράδοξο επίση να αυξήσουμε κάποιο σημαντικό τον ρόλο, την εντολή του Προέδρου ε, του διαχειριστικού, του, του διοικητικού οργάνου και ε, αυτό ωφελεί γιατί από την δική μου εμπειρία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δέλτα Νιτάφη ήμουν ο πρόεδρος. Όπως τώρα οι πρόεδροι αυτών των εποπτικών ε, συμβουλίων και οργάνων και θυμάμαι ότι το καταστατικό του Δέλτα μου έδινε το δικαίωμα να έχω την αποφασιστική κρίσιμη ψήφα αν υπήρχε ισοψηφία. Έτσι κι ήταν σπάνιες βέβαια ψηφορίες. Πολύ σπάνιες. Όμως αυτό περιβάλλει με ένα ιδιαίτερο κύριο στον πρόεδρο και το οποίο είναι καλή ιδέα. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την χρηματοδότηση, αυτό ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα. Σχετικά με του εθνικού προπολογισμού, να δούμε πώ θα υπάρξει αξιολόγηση και αναθεώρηση των σημερινών χρηματοδοτικών μοντέλων, οπότε και αυτό θα μπορούσε να γίνει λαμβάνοντας υπόψη της δημοσιονομικούς περιορισμούς για το ποιος είναι ο ρόλος της βιομηχανίας, το σχετικό μοντέλο χρηματοδότησης. Μόνο όμως εάν οι διαφορετικέ αρχές εμπλακούν σε άμεση εποπτεία, άπαξ και οι εισφορίες έχουν λόγο όσον αφορά τα χρήματά τους και το πώς αξιοποιούνται. Αλλά εδώ θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες επισημάνσεις και προειδοποίησεις στο σύστημα. Τώρα, για το πρόβλημα ή την πρόκληση του Brexit. Είναι και ευκαιρία ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε αναδιόριση και αξιολόγηση των εποπτικών αρχών του Ενωμένου Βασίλειου. Όντω είναι η βασική χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη και εκεί έχουμε συγκεντρωμένες δραστηριότητε των χρηματογόρων μας και μετά την αποχώρηση της Βρετανίας θα πρέπει 27 να θωρακίσουν τις αγορές τους. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα τα εξή. ότι θα πρέπει να περιοριστεί η κατάτμιση των αγορών που ισχύει σήμερα, γιατί γιατί δεν έχουμε οικονομίες κλίμακας και δεν έχουμε επίσης και αποτελέσματα δικτύου στους 27. 27 επίσης ίσως χρειάζονται να έχουν και υποπτικές λειτουργίες ε, άπαξ και έχουμε την μεταφορά αυτών των δραστηριοτήτων των αγορών από το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί μπορεί αυτό να γίνει σε σημαντικό βαθμό. Πώς να προχωρήσουμε. Ένα βήμα θα ήταν να προσδώσουμε σε αυτές τις εποπτικές αρχές το δικαίωμα να μπορούν να ενίστανται όσον αφορά τη χορήγηση κάποιων ε, εγκρίσεων ή αδειοδοτήσεων όπου εμπλέκονται μη αρμόδιες αρχές. Όποτε θεωρούν οι πολιτικές αρχές ότι αυτό είναι αντιστοιχεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άπαξ και έρθει το Brexit. Πρέπει 27 να είναι θωρακισμένοι ούτως ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν, να διατηρήσουν την ε, χρηματοπιστωτική τους ε, ακεραιότητα και τη συμμόρφωση προς τους κανόνες. Η ε, βασικό κέντρο παγκόσμιου ακτινοβολία. είχαμε πει ότι δεν έχουμε κάποια ρυθμιστική αρχή κάποτε ε, για αυτά και οπότε δεν υπήρχε. Αλλά είχαμε την Επιτροπή Χρημαστερίου, την SEC, τον ΙΠΑ που ήταν η, η μόνη ρυθμιστική αρχή όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σήμερα, βέβαια, αυτό το οποίο ακούω συνεχώς και διαλείπτως εδώ και 10-15 χρόνια, αυτό τώρα σταμάτησε να ακούγεται. Αλλά ίσως τώρα θα έχει σημασία ότι αυτή η Αμερικάνικη Επιτροπή Χρημαστηρίων να έρθει και στην Ευρώπη. Να έχουμε και εμεί τη δική μας δηλαδή SEC. Άρα είναι μια ιδέα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου το Brexit δεν μεταβάλλει την σημασία, την μεγάλη αυτών των υποπτικών αρχών. Αντιθέτως, η Ευρώπη χρειάζεται μια τέτοια αρχή ούτως ώστε να υπάρχει προστασία επενδυτών και CMU, οπότε θα πρέπει να αυξηθούν οι σχετικές αρμοδιότητες και των ε, διοικητών, των επικεφαλής αυτών των αρχών. Τώρα για την EBA είπαμε ότι έχουμε κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσες. Το Brexit θα έχει στην EBA άμεσες επιπτώσεις, μια που θα πρέπει να γίνει μετακόμιση από το Λονδίνο προς άλλη χώρα. Σε αυτή τη μικρή μου παρουσίαση δεν αναφέρθηκα σε αυτό που είπατε κύριε Πρόεδρε, το Twin Peak. Πάντως, όποιος έχει ερωτήσεις για το θέμα αυτό, ευχαριστώ να τις απαντήσω και εν κατακλείδη. Θέλω να πω ότι πέραν και ανεξαρτήτως του Brexit, Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τεχνικά πρότυπα μια αρχή για να υπάρχει η σύγκληση σε αυτά, για να έχουμε τα stress tests, για να υπάρχει η μεσολάβηση μεταξύ των χωρών όσον αφορά τα θέματα της εφαρμογής των αποκλήσεων. Είναι σημαντικό, θεωρώ, όχι μόνο να συνεχίσουμε να έχουμε τις ευρωπαϊκέ αρχές, αλλά και να τις αναβαθμίσουμε. Αυτό θα βοηθήσει όσον αφορά τη σύγκληση της εποπτείας στην ενιαία αγορά. Πολύ σημαντικό. Τώρα, για το μέλλον. Μετά τις διαπραγματεύσεις του Brexit, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα καθορίσουν τι σχέση θα είναι η πιο καλή, η πιο δόκιμη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένου Βασιλείου. Άρα τώρα δεν μπορούμε να προδικάσουμε ή να κάνουμε αξιολογικές κρίσει από αυτού. Όμως, να ολοκληρώσω με μια σκέψη μου. Νομίζω ότι, μια που είναι τόσο σημαντικό το χρηματιστήριο του Λονδίνου, θα ήταν προς το συμφέρον όλων ημών να χρησιμοποιήσουμε την ΕΣΜΑ ως μια πλατφόρμα μελούσης συνεργασίας. Και κατά την άποψή μου, στο πλαίσιο αυτό το να καταστεί το Ρωμανό Βασίλειο ρυθμιστής της αγοράς θα σημαίνει τροπεί του κανονισμού της ΕΣΜΑ. Καθεστώς παρατηρητή ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα. Και έτσι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξασφάλιζαν την ε, ευκαιρία να συνεργάζονται σε συντονισμένο με συντονισμένο τρόπο για τα σημαντικά αυτά θέματα. Και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια τέτοια αρχή στην Ευρώπη, η οποία θα φέρνει αποτελέσματα αυτή τη νέα η FCC όπως σας ανέφερα, θα πρέπει να μην διστάσουμε να την προωθήσουμε. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι και το Ρωμανό Βασίλειο και η ΕΣΜΑ θα έχουν θέση στο ε, διοικητικό της Συμβούλιο. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσπεπτη η ιδέα. Αφορά πάντως μόνο το μέλλον. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ρωμανό Βασίλειο θα μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για τα θέματα αυτά. Πάντως τα κρίνω σημαντικά. Και βέβαια μιλάμε μόνο για την διεθνή θεσμική συνεργασία το όντι, σημαντική, αλλά δεν πρέπει και να λησμονούμε πως ε, πέραν των θεσμικών ε, βελτιώσεων στις οποίες ανεφέρθην, δεν πρέπει να λησμονούμε τη βασική αρχή της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς την οποία χωρίς ένα βαθμό σύγκλησης σε θέματα οικονομικής πολιτικής, σε επιτεύγματα οικονομικής πολιτικής, θα είναι πολύ δύσκολο να πιεστούν χώρες σε θεσμικές βελτιώσεις, σε τήρηση των ουσιοδών εκείνων συνθήκων που διέπουν την εμπιστοσύνη. Και ειδικά σήμερα το ότι υπάρχει αυτή η κατακαιρματισμένη ε, τραπεζική ένωση που πόρο απέχει από το να είναι ένωση, οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη. Ας μην είμαστε λοιπόν υπερβολικά αισιόδοξε προς τις θεσμικές βελτιώσεις, σημαντικές πάντα, εφόσον βέβαια ε, προώθηθούν μετά από μελέτη και όριμη σκέψη, αλλά πιο σημαντικό θα είναι να ε, προωθηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών. Και σας ευχαριστώ. Κύριε Τιλαροζιέρ, σας ευχαριστώ και εγώ για, την πολύ σημαντική, για τις πολύ σημαντικές αυτές ε, ε, προτάσεις σας. πολύ σημαντικές και σκέψεις αλλά και ε, ανοίγματα, δυνατότητες δράσης. Ιδιαίτερα το τελευταίο που αναφέρατε για μια δυνατότητα, για μια πλατφόρμα συνεργασίας. Μου φαίνεται ιδιαίτερα φρόνιμη πρόταση. Ο Αλέλα Μασούρ είναι ο πρώτος ομιλητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τελαροζιέρ έχουμε μείνει εννοεί από τον τρόπο με τον οποίο παρακολούθησε την υλοποίηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τις συστάσεις της δικής του ομάδας του 2009 και βέβαια η δική του συνεισφορά είναι πολύτιμη για μας. Ε, έχω τις εξής ερωτήσεις για να αναφερθώ στην τελευταία από τις παρατηρήσεις σας κύριε Πρόεδρε. Στην έκθεση του 2009 εσείς εκφράζατε την ε, ευχή ούτως υπήν να υπάρξει μια ούτως υπήν αυθόρμητη αντίδραση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για να προχωρήσουμε σχεδόν αυτόματα ή αυθόρμητα σε μια ε, τραπεζική συνεργασία. Ταυτόχρονα λέγατε ότι κακώς παραμένουν παντοδύναμοι οι ε, νομοθέτες. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η αυτοματοποιημένη ενοποίηση της αγοράς και η Τραπεζική Ένωση είναι μόνο στα σπάργανα. Δηλαδή είχαμε μια αρχή, ελεύθερη αρχή ε, διαθέσιμη στη Βόρεια Ευρώπη, κάποιες απαρχές ακόμα και στην Ελλάδα ε, συνεργασίας, αλλά φαίνεται τελικά δεν επέτρεψαν οι εθνικές αρχές, επειδή δεν υπήρχε επαρκής ε, εμπιστοσύνη να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν θεωρείτε πως τα συστήματα εποπτείας, επαγρύπνησης ε, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην, στην θέσπιση αυτής της πραγματικής, της γνήσιας αγοράς ε, των εργασίων των ε, κεφαλαίων. Επίσης ε, μας ρίξατε το διπλό αυτό αγκίστρι. Ε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει άπαξ και η BA να αγκαστεί να αποχωρήσει από το Λονδίνο. Μήπως η ευκαιρία αυτή είναι χρυσή ευκαιρία για να αναμορφωθούν κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες ή πρέπει να μείνει το σύστημα όσο έχει. Παρακαλώ. Θα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και οι δύο αυτές ερωτήσεις συνιστούν μεγάλη πρόκληση. Η έκθεση λοιπόν ανάγεται στο 2009 όπου δεν είχαμε ακόμη διέλθει την κρίση των κρατικών χρεών του 2009, η οποία σώβησε τα χρόνια που ακολούθησαν. Λέτε ότι είχε εγγραφεί η έκθεση σε μια υπόθεση που έλεγε ότι μια ευρωπαϊκή ε, κεφαλαιοχική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπον αυθόρμητο θα δημιουργούνταν, δημιουργούνταν ε, όντως, όντως έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί ακολουθούσαμε την ιδέα ότι θα μπορούσε να ενοποιηθεί έτσι περαιτέρω από ό,τι είχε μέχρι τότε επιτύχει η κεφαλαιοχική χρηματοπιστωτική αγορά. Ωστόσο αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα ήταν ότι με την κρίση των κρατικών χρεών κατακαιρματίστηκε η αγορά διότι η εμπιστοσύνη, στην ε, οποία αναφερθήκαμε και νωρίτερα, έδωσε τη θέση της στην δυσπιστία. Και βέβαια αυτό είχε πολλαπλές συνέπειες. Συνέπεια καταρχάς για, τις, ε, για τους τραπεζικούς ομίλους, γιατί οι υπερσυνοριακοί τραπεζικοί όμιλη, και υπήρχαν κάποιοι ήδη το 2009, είχαν την ε, συνήθεια να θεωρούν εαυτούς ως ευρωπαϊκούς ομίλους που δεν ε, γνώριζαν σύνορα ή μελήματα ιδιαίτερα σχετικά με τις εθνικές εποπτικές αρχές στη διαχείριση των ε, ποθαματικών τους, της ε, ρευστότητάς τους και έτσι το 2009 ακόμα ε, εποφελούμενοι οι όμιλοι αυτοί από την ευκολία που τους έδινε η θεώρησή τους ως ομίλου προέβαιναν σε αυτή ακριβώς την επιλογή της χρηματοδότησης, δηλαδή ως ομίλου. Και υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι, οι οποίοι στη συνέχεια βέβαια διαλύθηκαν γιατί οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολικά μεγάλος ο κίνδυνος του να επαφίενται στην ε, φρονιμάδα αυτών των ομίλων και έτσι όρισαν ε, κανόνες ε, από θέματος ρευστότητας για τους ομίλους, πράγμα το οποίο δεν αντιστοιχούσε στις δικές τους επιλογές ε, για μια κεφαλο... κεφαλουχική αγορά διεθνή. Από την άλλη είχαμε και τις ε, αγορές οι οποίες έδειξαν μεγάλη μεγάλο φόβο εναντί των ε, spread, των μεγάλων αποκλήσεων και έτσι οδήγησαν σε κατακαιρματισμό των ε, ε, κεφαλαίων. Έτσι λοιπόν σωστά μας λέτε ότι το έχουμε το οικονομικό σύστημα το οποίο έπρεπε να είναι το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι λειτουργεί ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Είναι ένα σύστημα που πρέπει να είναι ενοποιημένο μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όμως δεν είναι ενοποιημένο. Τουναντίον είναι πολύ πιο κατακαιρματισμένο από ό,τι θα έπρεπε. Έχω μάλιστα συντάξει υπόμνημα μαζί με άλλους ε, οικονομολόγους το 2012 συγκεκριμένα ως προς την αδύρυτη ανάγκη, εφόσον βεβαίως θέλουμε μια ε, τραπεζική ένωση έτσι μάλλον ε, κεφαλαιακή ένωση, να εξασφαλιστεί δυνατότητα κινητικότητας των ε, κεφαλαίων, δηλαδή να μπορούν να πηγαίνουν εκεί όπου βλέπουν πως υπάρχουν δυνατότητες για επενδύσεις. Για άλλη μια φορά λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό και ενδιαφέρον. Δεν πρόκειται ε, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις ε, της ευρωπαϊκής πλευράς να επιτρέψουν την ε, ανάκτηση αυτής της εμπιστοσύνης ή την απόκτηση αυτής της εμπιστοσύνης μόνο με ε, μέτρα εξασφάλισης εμπιστοσύνης θα μπορέσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Για το διπλό αγγίση, το Twin Peak, ε, έχω κάνει τη σχετική μου μελέτη με πειράματα που έχουν γίνει μάλιστα και στο παρελθόν σε σχέση με την ε, ανάθεση στον ίδιο φορέα και της επαλήθευσης και του ελέγχου για τις τράπεζες Φερρυπίν και υπάρχουν ε, κάποια πειράματα που έφεραν καλά αποτελέσματα, κάποια που ήταν λιγότερο θετικά. Σε τελευταία ανάλυση τα πάντα εξαρτώνται από το περιβάλλον και από την οτροπία των ε, επικεφαλής ε, αυτών των οργανισμών. Έτσι λοιπόν δεν θα έλεγα εύκολα ότι είναι μια πολύ καλή λύση που ε, ρυθμίζει τα προβλήματα. Δεν θα τολμούσα να το πω αυτό και εν αμφιβόλω μάλιστα θα έλεγα ας μείνουμε καλύτερα μακριά. Θα έπρεπε να υπάρχουν ίσως λόγοι σοβαροί για να το πράξουμε δεν είμαι πεπισμένο ότι συγκεντρώνονται αυτοί οι λόγοι. Ευχαριστώ, Περβάνος πέχές Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Οικονομική Νοσηματική Επιτροπή. Συζητούμε το θέμα αυτό και θεωρώ ότι έπρεπε να συζητήσουμε μαζί σας διότι το καθεστώς το οποίο ζούμε οφείλει πολλά στις εκθέσεις που εκπονήσατε εσείς με πολλές ε, συζητήσεις με αυτό το κοινοβούλιο. Έχω δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στο θέμα της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτή η Τραπεζική Ένωση προσετέθη στο μηχανισμό ΣΕΖΑ που υπήρχε. Τροποποιήθηκε κάπως ο μηχανισμός θεσπίζοντας ένα νέο φορέα, το ΣΕΣΕΜ. Θεωρείτε ότι αυτά, αυτό αλλάζει τα δεδομένα. το αναφέρατε ακροθυγό στα πλαίσια του ΕΣΜΑ κατά κάποιο τρόπο μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο για το ΕΣΜΑ και το ΕΟΠΑ. Άλλη ερώτηση. Αναφερθήκατε στον κατακαιρματισμό που συνδέεται με την κρίση του κρατικού χρέους που ξύπνησαν οι οίκοι αξιολόγησης κλπ. Όλα αυτά που ζήσαμε τέλος πάντων όλα αυτά κατέστρεψαν τη δυναμική των τραπεζικών ε, ομίλων των διεθνών. Και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την κατάσταση ε, μέσω ενός ενιαίου εχειριδίου κανόνων και σταδιακά οι εποπτικές αρχές ε, θα κινηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της, της διεθνούς αυτής ομάδας που υπάρχει και ότι είναι ενδιαφέρον να έχουμε τους θεσμούς ε, για να μπορούμε να λειτουργούμε αποτελεσματικότερα όσον αφορά την αγορά κεφαλαίων στην Ευρώπη. Μήπως στάσαμε σε ένα στάδιο που θα πρέπει να επανέλθει η ιδέα το 28-21 το καθεστώς, ειδικό καθεστώς για τις μεγάλες ε, υπερεθνικές τράπεζες. Και τρίτη ερώτηση. Δεν μπορώ να αντισταθώ, βλέπετε βασιζόμενοι σε αυτά που έλεγε ένα Μασούρ, το φαινόμενο Twin Peaks. Όταν μιλάμε για Twin Peaks, σκεφτόμαστε το παλιό Ολλανδικό μοντέλο των ασφαλιστικών τραπεζών. Μιλάμε για άλλη τάξη μεγέθους τώρα. Ε, ποιο, είναι θα δυνατότητα προσεγγίσεως των συστημάτων ε, της Ευρωπαϊκής Τραπεζική Αρχής με το σύστημα SSM, εμπα SSM. Αγαπητή Περβάν ε, Περέζ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σου. Η πρώτη ερώτηση, σημαντικότατη, αφορά την όλη δομή. Δηλαδή, είπατε σχεδιάσατε το σύστημα το 2009, είχε μια λογική το σύστημα τότε και όταν δημιουργήσαμε τραπεζική ένωση κάποια χρόνια μετά, οι δύο λογικές που ακολουθήθηκαν δεν συνέπιπταν άριστα και δεν συγκατοικούν πολύ καλά. Είναι ένα θέμα που με απασχόλησε και εμένα τότε. Η απάντησή μου είναι εξή. Αυτήν έδινα πάντα όταν με ρωτούσαν. Έλεγα και λέω. Η δημιουργία του SSM που όλες οι χώρες της Νομισματικής Ένωσης το χρησιμοποιούν σαν μηχανισμό τον εποπτικό τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Δεν νομίζω λοιπόν η δημιουργία αυτού του συστήματος, του SSM, αλλάζει επουδενή τη λογική, τη βάσιμη λογική της ε, ΕΜΠΑ. Γιατί το λέω αυτό. Το SSM δεν είναι ρυθμιστικός φορέας. Είναι σημαντικότατο να σημειωθεί αυτό. Ακολουθεί την προσέγγιση η Λαμφαλουσή, πρώτο, δεύτερο, τρίτο επίπεδο και εφαρμόζεται όχι μόνο στα μέλη της ΟΝΕ και τις υποψήφιες χώρες συμμετοχή στο μηχανισμό, ο κανονισμός, η όλη ρύθμιση εντάσσεται πάντα στον τομέα της ΕΜΠΑ. Αν καταργούσαμε την ΕΜΠΑ διότι θα επικρατούσε, θα υπερίσχυε το SSM, τότε θα χάναμε το Common Rule Book. Ποια είναι η εμπειρία μου, ότι χωρίς το Common Rule Book δεν υπάρχει ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά. Πρέπει να διαφυλαχθεί. Βέβαια, χρειάζεται να προσαρμοστεί η ΕΜΠΑ με τη μεσετοχή των μελών της ΟΝΕ και όσον αφορά τον τρόπο ψηφοφορίας λάβαμε υπόψη τις σχετικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ίσως τώρα δεν είμαστε στο ίδιο γεωγραφικό πλαίσιο πλέον με το Brexit πρέπει να επαναξεταστεί το ζήτημα των κανόνων ψηφοφορίας που είναι περίπλοκη. Το άλλο ερώτημα που θέσατε. του 28ου καθεστώτος. Πιστεύω ή θα έτεινα να πιστεύω δεν το σκέφτηκα αρκετά το ερώτημα που θέσατε. Εγώ τίνω να πιστεύω ότι το 28-8 καθεστώς ε, είναι ένα καθεστώς με δυνητική εφαρμογή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του καλύτερου καθεστώτος και αυτό κάπως αν το κάνουμε όμως ε, θα απαρνηθούμε κάπως στον 9 αγορά δεν θέλουμε 27 καθεστώτα και να προσχωρήσει ένα 28 καθεστώς. Ε, η έννοια που αντιλαμβάνομαι είναι να έχουμε ένα κοινό καθεστώς του Common Rule Book. Είναι δογματική απάντησή μου, αλλά προς τα εκεί κινούμε. Για το Twin Peak. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Στις Ηνωμένε Πολιτείες, εδώ και κάποιες μέρες, μεγάλος Αμερικανός, ο Πολ Βόκερ, που σέβεται όλους, είπε ότι ήταν παράλογο να υπάρχουν έξι οργανισμοί ελέγχου όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά. Διότι είναι έξι. Η Fed, ο FDSC, Control of Currency, οι αρχές οι πολιτιακές για την ασφάλεια, για την ασφάλιση και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι. Δεν είναι Twin Peaks. Είναι μεγάλος ο διαχωρισμός και κατακαιρματισμός. Εμείς καλά τα καταφέραμε θα έλεγα. Έχουμε τρία peaks. Έχουμε τις ασφαλείς, τις ασφάλειες, τις τράπεζες και τη χρηματοσυντητική αγορά. Προφανώς ε, το ένα επισύρχεται στο άλλο. Και μπορούμε να πούμε ότι το καλύτερο οικοδόμημα θα ήταν ε, να καλύψουμε χρηματιστικές αγορές, τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες ε, με μία κίνηση. Προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτές οι θεσμικές ενοποίησεις οδηγούν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας. Δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω ότι ο κόσμος ασφαλιστικός διαφέρει πολύ από τον τραπεζικό. Δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Δεν είναι τα ίδια δημοσιο... χρηματοπιστωτικά σαν προσεγγίσεις. Πιστεύω ότι άλλο οι τράπεζες, άλλο οι ασφαλιστικές εταιρείες, ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, κάτι άλλο. Μπορούμε να δείξουμε ότι με ενιαίο φορέα είμαστε πιο καλά τρόφο ε, καλυμμένοι και δημιουργούνται συμπράξεις και μια συμβίωση των φορέων. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Είμαι αρκετά διστακτικός όσον αφορά αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε αυτό που συχνά γίνεται στην Ευρώπη, υπάρχει τόσο πειρασμός, να τις θεσμικές αλλαγές να τις ε, χρησιμοποιούμε σαν ε, φωτεινό οδηγό. Έχουμε μόλις ένα δεκάλεπτο. Ας ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις και μετά θα σας δώσουμε το λόγο στο τέλος. Κέι, θέλεις να πεις κάτι? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, η αρχική σας δουλειά έγινε πριν από χρόνια, το μεταξύ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν για την, ε, μετα... για την περίοδο μετά την οικονομική κρίση και βέβαια θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι ανεγνωρισμένη η δουλειά σας. Ταυτόχρονα υπάρχει και άλλος τομέας στον οποίο σημειώθηκε σημαντική πρόοδος που είναι η παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ε, ε, εποπτών και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό να υλοποιείται, ωστόσο το σύστημα δεν λειτουργεί πάντα ικανοποιητικά, όπως η παραδείγματι στην ε, αναγνώριση των εποπτικών αρχών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Όταν λοιπόν ηγείται τέτοιων ε, αναγνωρίσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε να πηγαίνει σχετικά καλά η κατάσταση. Όταν όμως έχουμε εθνικές αρχές ε, πολύ πιο δύσκολα φέρνει αποτελέσματα το σύστημα και ξέρω ότι η δυσφορία εκφράζεται και στον Καναδά και την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες δικαιοδοσίες. Ένα τέτοιο λοιπόν τεχνικό χάσμα θα έπρεπε να καλυφθεί για το μέλλον. Βλέπετε κάποιους ε, φραγμούς ε, θεσμικούς ενδεχομένως και θα μπορούσε για το μέλλον η ΕΣΜΑ να αναλάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις και κινήσεις στο μέλλον αντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερώτηση, ε, απάντηση, καλή ερώτηση, λέει ο κύριος Πολιτιέρη, για να δούμε αν υπάρχουν άλλοι. Κύριος Λαμασούρ, για άλλη μία. Ναι, σε συμπλήρωση της ερώτησης που ακούσαμε, και μια και έχουμε τον Ζάκλα Ροζιέρ εδώ που έχει τεράστια εμπειρία θα ρωτήσω το εξή, ότι δεν έχουμε ακόμη αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εκπροσώπησης ούτε στο Δουνοτού ούτε και σε άλλους ε, χρηματοοικονομικούς, χρηματοπιστωτικούς φορείς ε, της ζώνης του ευρώ. Αυτό το πρόβλημα πώς θα μπορούσε να λυθεί. Ευχαριστώ, Τάν. Ναι, Πρόεδρε, σύντομα, κατά το δυνατόν και ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σας και η ομιλία σας. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέζει προς μια ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κεφαλαιακών αγορών με αρκετή υποστήριξη εδώ στο Κοινοβούλιο. Από την άλλη πρέπει να πω ότι ε, με έκπληξη διαπιστώνω πως ε, δεν αναφέρεται στις σχετικές προτεραιότητες η ευρωπαϊκή εποπτεία. Θα σας καταλαβαίνω καλά από τα όσα είπατε ότι θα θεωρούσατε σκόπιμο να υπάρχει αυτό και ότι θα έτεινε προς τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κεφαλαϊκής αγοράς και εν πάση περιπτώσει τι θα θέλατε να δείτε σαν ε, ε, απάντηση, τι θα έπρεπε ακόμα να γίνει. Το Brexit μου φαίνεται, μου να το χαρακτηρίσατε με τα λόγια σας ως ευκαιρία αλλά ταυτόχρονα είναι και μία απειλή η JP Morgan φεύγει από το Λονδίνο για να περάσει τις δραστηριότητες της στην Ευρωπαϊκή χώρα είναι και απειλή μαζί μπορεί να οδηγήσει σε κατακαιρματισμό για την ίδια την ε, υπηρετική Ευρώπη εάν αυτές τις δραστηριότητες προσπαθήσει κάθε κυβέρνηση για λογαριασμό της να τις ε, προσελκύσει ο, ο πρόεδρε ευχαριστώ πολύ για το πρώτο θέμα της συνεργασίας για, μεταξύ των σημαντικών παγκοσμίω δικαιοδοσιών. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει αναλάβει ηγετική δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα στη διαπραγμάτευση του ζητήματος των ισοδυνάμων που βεβαίως ε, ε, οδηγεί σε δυσφορία άλλες αρχές που έχουν συνηθίσει να έχουν αυτόνομη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. Όντως, πρόκειται για ένα ζήτημα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι την κατάσταση ως εξή. Όσο δεν είμαστε μια απολύτως γνήσια ένωση, ένωση δηλαδή όχι κρατών μελών, όπως τώρα, ε, παραμένει λογικό να είναι η Επιτροπή εκείνη η οποία θα αποφασίζει για τέτοια ζητήματα όπως οι ισοδυναμίες. Γιατί εάν αυτά τα αναθέσουμε σε εποπτικές αρχές, χάνουμε τη πολιτική βαρύτητα της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή είναι περισσότερο θα έλεγα εκπρόσωπος του, ε, της Ένωσης από ότι θα, θα ήταν η ΕΣΑ Φερρυπίν. Τώρα αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο θα διευκρινιστούν ζητήματα των αντιπροσωπιών ε, αλλά πάλι καταλαβαίνω όλες τις ε, ε, παρατηρήσεις και την ε, δυσφορία για τον κύριο Λαμανσούρ, που αναφέρθηκε στην εκπροσώπηση της Ένωσης σε σώματα όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μα θα του δώσω την ίδια απάντηση. σου έχουμε την αίσθηση ότι τα συμφέροντα της Γαλλίας στην συζήτηση ενός μελλοντικού διεθνούς συστήματος εποπτείας είναι τόσο σημαντικά και είναι τόσο ιδιαίτερα που δεν μπορούν να στηριχθούν σε έναν φορέα που θα εκπροσωπεί την Ένωση. Όσο έχουμε αυτή την οτροπία δεν θα υπάρξει εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Δούνο του στο Διοικητικό σύμβουλο του ΔΝΤ Γιατί ακόμη δεν έχουμε οικοδομήσει αυτήν την κοινότητα συμφέροντος, τα λοιπά, που θα ήταν αναγκαία και επαρκής. Και έτσι... Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να δράσουμε ως χώρα για να μπορέσουμε να έχουμε την εκπροσώπωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δουνουτού ή του Παγκόσμιας Τράπεζας. Επίσης, θα συμπληρώσω ότι με το Brexit θα έχουμε ε, αν, αναπόφευκτα αλλαγές ως προς τις έδρες χρηματοοικονομικών οργανισμών της Ευρώπης. Αλλαγές οι οποίες εξορισμού θα τείνουν προς περισσότερες μετατοπίσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την υπηρετική Ευρώπη. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει, αντίστροφα δεν μπορεί να γίνει. Τι θα φέρουνε, δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι μεγέθη θα κινηθούν αυτές οι αλλαγές, πάντως δεν θα ξεφνιζόμουν, αν ήταν αρκετά μεγάλο όγκου. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε εμείς εδώ στην υπηρετική Ευρώπη και να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν πιο ε, πιδέξια, ασφαλή ως προς την νομοθεσία, ενωτική συμπεριφορά με κανόνες, με φορείς, ε, ε, δηλαδή να, είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάμε καλά, ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα αντέξουμε. Και ότι θα είμαστε τουλάχιστον εισάξιοι με, το, με τα σχετικά όργανα υποπτίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, σας έδωσα μερικά παραδείγματα του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τη διευκόλυνση της υλοποίησης αυτής της ε, διευρυμένης ε, νομισματικής, ε, χρηματο, χρηματονομισματικής ένωσης, χρηματοπιστωτικής ένωσης, πάντως ήταν μεγάλη πρόκληση. Πάντως φρονώ ότι δεν πρέπει να λησμονήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση της ε, χρηματοοικονομικής αγοράς μετά το Brexit. Και να έχουμε μια χείρα συνεργασίας απλωμένη προς τους Βρετανούς και να τους πούμε δεν είναι προς το συμφέρον όλων μας να οργανώσουμε τα πράγματα κατά τρόπο συνεργατικό και όχι χαοτικό. και επίση αναφέρθηκε στα CCP. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Όχι, καλώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ήταν εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων. Θα μελετήσουμε, θα αναλογιστούμε τα θέματα αυτά που μας εκθέσατε συμπεριλαμβανομένων και των επιφυλάξεων σας για τις ε, δικέφαλες αρχές. Όπως και να έχει θα κοιτάξουμε την, ε, τις προοπτικές για τη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ενιαίας ε, αγοράς για το χρηματοοικονομικό τομέα και βέβαια την δυνατότητα λειτουργίας μιας πραγματικής εποπτικής αρχής. Σας ευχαριστώ. Yeah, he said I should. He don't. Dear colleagues, if we can continue to make sure that we will start voting on. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία το ταχύτερο. Έχουμε τον ΦΠΑ στα βιβλία καταρχάς. Με τον Τόμ, αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να σας τα πω ή στα Ολλανδικά, εάν δεν έχετε πρόβλημα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί ήταν πολύ επικοδομητικές οι τροπολογίες τους. Ε, βέβαια έτσι μπήκα σε πειρασμό, αλλά το κείμενο ήταν κάτι το οποίο επιβάλλεται να γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω τώρα. Γιατί στο καλό δεν το κάναμε νωρίτερα. Να, ένα παράδειγμα όμως το πώς η Ευρώπη μπορεί να κάνει πράγματα που να αγγίζουν τον κόσμο. Υπήρχε άνηση μεταχείριση. Έπρεπε αυτό να ρυθμιστεί. Οπότε είπαμε για ευελιξία προ τα κατημέλη, ούτω να κανονίσουν του συντελεστέ τους. Εγώ πρότεινα μια συμβαστική τροπολογία για να καλύψω του συναδέλφου. και να καλύψω και την πολιτιστική μας επιτροπή. Ελπίζω δεν υπάρχουν προβλήματα. Όπω δεν υπήρχαν προηγουμένω και στην ε, ψήφιση. Ευχαριστώ του σκιώδει ηγητέ. Ήταν πολύ επικοδομητική η θέση του. Έχουμε από του σοσιαλιστέ σκιώδη ηγητή, ρωτά ο πρόεδρο. Α, η κυρία Μπερέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ η συνάδελφο. Αλλά ανταυτή, εγώ θα σα πω τι θέλει. Θεωρεί ότι η, η έκθεση δεν παρουσιάζει προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάποιες προτάσεις ε, κρυστάλλινες και τα έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρα ο εισηγητής και με τις τροπολογίες. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτό το οποίο ισχύουν τώρα όσον αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία και ο συντελεστής ε, επίσης για για τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και πολλα κρατημέλη ήδη εφαρμόζουν μειωμένους ή υπερβολικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΒΠΑ ή κάποια βιβλία ως πολιτιστικό προ... Μα γιατί πάντα εγώ λαμβάνω το λόγο όταν οι άλλοι ετοιμάζονται να ε, προσθέτουν την ψηφοφορία. Παρακαλώ κάντε ησυχία γιατί μιλούμε για το θέμα πριν την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε θέσπισαν πάνω από 50% τον κλασικό συντελεστή για τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, τα ελληνικά περιοδικά κλπ. Και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή είναι η τεχνολογία. Δεν αλλάζει το περιεχόμενο στην ουσία του ε, και επίσης έχουμε καινοτομία τώρα για αυτές τις δημοσιεύσεις. Θέλαμε να είναι η έκθεση όσο γίνεται πιο ευσύνοπτη, πιο ξεκάθαρη και να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα στο Συμβούλιο ότι αυτή η πρόταση πρέπει να υφετηθεί το συντομότερο δυνατόν. Και για αυτό και δεν κατεβάσαμε εμείς τροπολογίες, αλλά είμαστε υπέρ των τροπολογιών που συγκλίνουν προς αυτά που είπα προηγουμένως, την καινοτομία ας πούμε και τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Δίνεται αυτή η έμφαση και αναδεικνύει ακριβώ αυτές τι πτυχές. Τροπολογίες 3 και 4, εντάξει, όσον αφορά τον, τη διάκριση μεταξύ αυτής της πρότασης και το άλλο πιο περίπλοκο θέμα της γενικότερης, ευρύτερης εναρμόνισης των συντελεστών φι, πι, α. Ε, γι' αυτό και εκεί που ζητεί περισσότερη ευελιξία από τα κράτη-μέλη δεν μπορώ να συμφωνήσω. Εκεί που λέει για μειωμένους συντελεστές αλλά θέλουμε να υπάρχει η κοινή λίστα με μειωμένο συντελεστή. Δεν συμφωνούμε με εκείνες τις τροπολογίες που αποδυναμώνουν την πρόταση. Και δεν είναι εκτός θέματος. Τώρα, σύμφωνα με το τι θα κάνουμε για την τροπολογία της Άλτε. Αναλόγως λοιπόν μπορούμε κάτι να προσθέσουμε για τον ορισμό. Τούτο σημαίνει για μας ότι εμένουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Μπερές. Ο Μπέντ Λούκα από την ECR, όχι, καλύτερη πίεση ο χρόνος, για κόρα από την Αλντέ. Παρακαλώ ένα λεπτό στα Ολλανδικά. Ναι, ναι, ναι. Εθ και εγώ θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα όπως μίλησε και ο στα Ολλανδικά. Θέλω να τον συγχαρώ γιατί είναι ευσύνοπτη αυτή η έκθεση. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Από πλευρά Άλντε, εμεί αυτό το ζητούσαμε να υπάρχει ε, ισότιμη μεταχείριση ε, μεταξύ βιβλίων και ηλεκτρικών βιβλίων. Οπότε το συντομότερο που θα το δικαιπεραιώσουμε το καλύτερο. Ο πρόεδρο, ευχαριστούμε. Πινελόπι Μπερμέχο της Γκουε είναι εδώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα όλα τα θέματα να είναι το ίδιο απλά όπως αυτό. Γιατί αυτό που δεν μπορώ να καταλαβώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έκανε αυτή τη διάκριση μεταξύ εφημερίδων, περιοδικών, ανάλογα αν ήταν σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Πάντοτε θα πρέπει ο σκοπός να είναι η εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό, στην κουλτούρα και να υπάρχει επίση ε, ποιοτική απασχόληση. Οπότε γι' αυτό και εγώ σα επισημαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε το ότι δημόσια κέντρα έρευνας να έχουν πρόσβαση σε υλικό πολιτιστικό χωρίς τροχοπέδες ε, φορολογικές όπως ίσχυε. Έχουμε τρόλες αυτές τις εκθέσεις για τον ΦΠΑ, άρα θα πρέπει να επιλέξουμε κατά πόσο θέλουμε να υπάρχει ένας τέτοιος εισπρακτικός μηχανισμός, ο οποίος θα είναι μη προοδευτικός και φύγει τις ε, πιο στοιχειώδεις ε, υπηρεσίες και κοινωνικά δικαιώματα σε σχέση με τον πολιτισμό ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φορολογία ούτως ώστε να δώσουμε αντικίνητρα για την κατανάλωση πολυτελείας. Άρα θα πρέπει και στο μέλλον να έχουμε την ίδια συνένεση όπως και σήμερα. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κάποιος από τους Πρασίνους. Όχι. Βλέπω όμως την Μπάρμπαρα Κάπελ. Μήπως δεν είναι... Α, εδώ είναι, εδώ είναι. Έχεις το λόγο. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρόκειται όντω για ένα τομέα στον οποίο πραγματικά μας μένει η απορία γιατί οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται με το ποσοστό, με το στελεστή του μειωμένου, στελεστή ΦΠΑ στα κράτη-μέλη μεταξύ των κρατών μελών ε, πρέπει να έχει ε, προχωρήσει αυτή η υπόθεση, κάτω από το 5% δηλαδή ΦΠΑ. Ωστόσο θέλω να σημειώσω ότι η πρόταση, όπως έχει εδώ, για την αλλαγή του συνήθους φορολογικού συντελεστή για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή ε, και θέλω επίσης να πω ότι για την επόμενη συνεδρίαση καλό θα ήταν να ε, προβλέψουμε και το ε, περιεχόμενο το μουσικό ή βίντεο. Γιατί και εδώ μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε την ε, δημιουργική, το δημιουργικό κλάδο, την πνευματική δημιουργία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είμαστε στην ώρα να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία. Παρακαλώ τον Μάρκους να φροντίσει για αυτό το θέμα. So, okay everybody, we start with the... Καλώς ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Έκον, έκον μόνο. Μόνο μέλη της έκον δικαιούνται για να ψηφίζουν. A test on Econ. Δοκιμή πρώτα παρακαλώ. Μέλη της έκον μόνο. Who is taking care here? And, and then is safeguarded that leader is not voting? This too much, Well, we are dependent from technique. That is uh, not a pool position. okay, I close the vote. Λοιπόν, ωραία, είδαμε ότι δουλεύει η τεχνολογία ικανοποιητικά. Σίγουρα εγγυημένο ότι είναι μόνο δισεκον. Ωραία, τροπολογίε υπέρ, 5 υπερ αποχέ. Ε, απορρίπτεται 6 υπερ Απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται 24 υπέρ κατά. Α επαληθεύσουμε, αν και μου φαίνεται ότι έχει εγκριθεί. Και άρχεται η ψηφοφορία. 24. Ψηφίσατε όλοι. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Αδιανόητον. Έναν αναπληρωτή, αναπληρωτή παρακαλώ. Τον έχετε. Μα δεν σας μετράμε καν γιατί δεν ανήκετε στην Επιτροπή. Καλά. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Ε, δεν ήταν και τόσο σαφέ. τελικά. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 συμβατή κατά αποχές απερίφθη, 1 κατά αποχές εγκρίνεται κουλτ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2, 3 ε, της κουλτ υπέρ κατά εγκρίνεται 14 υπερκατά. Κύριε Λάγκη, είναι σοβαρή η Ε, αποχές εγκρίνεται 15 Τι υπέρ ήσασταν 14. Καλά, ε, επαληθεύουμε τη 14. η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι και πέρας. Και όντω εγκρίνεται. συγγνώμη. Να σέβεστε τον πρόεδρο, να εμπιστεύεστε τον πρόεδρο ακόμα και αν δεν είναι τη ομάδα σα. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία, 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, κουλτ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ονομαστικά πέρας. Ψηφίσατε όλοι. Περισσεύουν τέσσερις του ΕΛΚ. Και ένας του Άλντε. Ε, όχι συναδελφοί, είμαστε πάντα στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Άλλο αυτό τώρα, άσχετο. Πρώτα μόνο η έκον για την ονομαστική, η οποία είναι επικίνδυνη για ορισμένους. Ε, ψηφίσατε όλοι λοιπόν, ωραία. Ο Ιάκοπ Φον Βάιτσεκερ έχει μια ακόμη ψήφο γιατί δεν είχε την κάρτα του. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αγαπητέ, ο κύριος Λάμπερτς, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Είμαι λίγο σαν τον Ιάκοπ Φον Βάιτσεκερ σήμερα. Μπορεί να είναι ψηλό αυτός και εγώ κοντός, αλλά... Και εγώ λησμόνισα την κάρτα μου. Oh. Κακό παιδί ακούγεται μέσα από την αίθουσα. Ξέρετε, κανονικά όταν προεδρεύω εγώ, κάτι τέτοια δεν τα επιτρέπω. Και η ε, θα με ψέξει αν το δεχθώ εκ μέρου σα. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Αν το δεχθήκατε για έναν ψηλό Γερμανό, δεχθείτε το και από έναν κοντό Βέλγο. Ναι, όχι, το δέχομαι γιατί φοράς κόκκινη γραβάτα. Μα άλλον δεν έχω δώσει το λόγο. Εντάξει, τέλος της συνεδρίασης της ΕΚΟΝ. Ανακοινώσεις άλλες, ε, προσεχή συνεδρίαση γνωστή και πέρα στη συνεδριάσεως.